Ladies and gentlemen, good afternoon. Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Πρέπει να έχετε μπροστά σας το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Πριν εγκριθεί, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ότι μεταδιδόμαστε στην ιστοσελίδα και θα σας χορηγηθεί και ένα βιβλιαρίδιο που λέει πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι όλοι ικανοποιημένοι από την ημερήσια διάταξη, αν ναι, τότε εγκρίνεται και περνάμε στην έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων. Εάν τεθεί καμία αντίρρηση να φανεί αμέσως όχι, ευχαριστώ πολύ, εγκρίνονται και αυτά. Επόμενο θέμα, διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου απολυμμένες. Θα, θα εξεταστούν οι τροπολογίες από τον εισηγητή κύριο Στέρκος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει τροπολογίες. Πιστεύω ότι ε, τα έγγραφα αυτά νομίζω ότι συμφωνούν με το γενικό πνεύμα. Σε μερικά σημεία θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζουμε όλοι ότι απαιτείται μία απλοποίηση διοικητική κατά τον κατάπλου από πόπλου. Εντάξει, αυτά συμφωνούν όλοι. Και μετά θα πούμε μερικά πράγματα λεπτομερέστερα. Πρόεδρε, θα ήθελα να αφαιρθώ για ορισμένα σημεία, όπως χάρη το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστούμε τον Μαρινέσκου για τις τροπολογίες που έχει υποβάλει αλλά στον κατάλογο ψηφοφορίας δεν τα έχω αυτά γιατί δεν νομίζω να χρειάζονται παρόμοιες τροπολογίες. Άρα λοιπόν ε, δεν τις με αυτές τις τροπολογίες και επειδή αναφέρει ότι ε, το πλοίο παραμένει στο λιμένα είτε τα πολεμικά πλοία τα οποία αποκλείονται ναι. από το πεδίο εφαρμογή αυτό εδώ. Δεύτερο σημείο τώρα είχα υποβάλει την τροπολογία 15 για την ηλεκτρονική δήλωση. Θέλουμε με την τροπολογία αυτή ε, να διευκρινίσουμε ότι ένα φαξ δεν είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γιατί χρειάζεται ακόμη μια κάποια επεξεργασία από το φαξ για να καταλήξει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα κείμενο και το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, αποτελεί ένα πολύ σωστό ορισμό. Και το κείμενο είναι καλύτερα από τις τροπολογίες Βλάστο και στην αρχή έλεγα να αποσύρω τη δική μου και να θετήσω του συναδέλφου, αλλά τελικά μου φαίνεται η δική μου τροπολογία ότι είναι καλύτερη. Και ακόμα το άρθρο 5, γλώσσα. Εκεί είναι αρκετά ριζοσπαστική η τροπολογία μου. Μία και μόνο γλώσσα, αγγλικά και με την Ισπανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήλθα άτυπα σε επαφή και το Συμβούλιο μου είπε άνοιχτα ότι το θέμα αυτό θα ήταν ιδιαίτερα λεπτό και δύσκολο. Καταλαβαίνω βέβαια πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εύκολο για μια γλώσσα για τα αγγλικά, αλλά στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επιτευχθεί μια γενική συμφωνία από τους περισσότερους για να θετηθεί μία και μόνο γλώσσα. Μετά τι θα κάνουμε όσον αφορά τη διατύπωση, δεν το ξέρω. Αλλά παρακαλώ συνάδελφοι να απορρίψετε τις πολυπιτροπολογίες και να υποστηρίξετε τη δική μου. Μετά, εκ των υστέρων, θα δούμε το αποτέλεσμα αυτό, το ευκταίο, πώς θα το πετύχουμε και θα ζητήσω παντός, ζητάω από τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών να υιοθετήσουν μια σαφή και συγκεκριμένη θέση και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και αναθετήσουμε μια περισσότερο ριζοσπαστική θέση. Το επόμενο σημείο που είναι το άρθρο 7, τρία πράγματα θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Πρώτα απ' όλα την ημερομηνία θέση σε ισχύ. Και ακόμα την επιλογή πλατφόρμας για τους υπολογιστές. Τι ακριβώς θα γίνει πώς θα γίνει η διαχείριση των στοιχείων ανάλογα με τις ανάγκες κλπ. και μετά πώς θα ανταλλάσσονται αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να μας εξηγήσει η Επιτροπή γιατί αναφέρει για μια σημαντική έτσι, ε, ημερομηνία. Εμείς δεν ασχολούμεθα μόνο με αυτό το θέμα ε, πολλές και διάφορες ρυθμίσεις ε, χάρη σε τελωνιακά θέματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι για αυτό το 2013. Γιατί να μην πάμε στο 2015 παραδείγματος Αυτό χρειάζεται να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο και θα πρέπει να προβάλλουμε και εμείς τα επιχειρήματά μας ότι όσο ταχύτερε πετύχουμε την απλοποίηση τόσο καλύτερο θα είναι. Δεν νομίζω να συμφωνήσουν όλοι, αλλά υπάρχουν σε άλλες ρυθμίσεις από τη Μουλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες πτυχές που έχουν ρυθμιστεί και θα πρέπει να τα δούμε, να τα δούμε και αυτά εδώ και να προχωρήσουμε σε ένα συντονισμό όλων. Γι' αυτό για την ημερομηνία να ισχύσει τελικά αυτό το 2013 και επίσης διάφορες τροπολογίες ε, υπέβαλα για το σύστημα των υπολογιστών, πώς θα αναφέρεται, πώς θα εξηγείτε. και από το Συμβούλιο τι μου υπόθηκε δεν θα είναι πια το safety το κύριο θέμα, το κυρίαρχο σύστημα, γιατί είναι αρκετοί που δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν αυτό το σύστημα. Αλλά λοιπόν πάνω σε αυτό το σύστημα θα πρέπει να το αναλύσουμε καλύτερα αυτό και επίσης 52-54 τροπολογίες και την πρόσβαση στα στοιχεία. Εγώ προχώρησα στη σύνταξη μιας ε, συμβιβαστικής λύσης η οποία συμπεριλαμβάνει την ε, τροπολογία Βλάστο, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της και μετά μιλάνε και καντράουι στις τροπολογίες τους που αναφέρεται από την αιτιολογική σκέψη και μετά. Και μετά η ιδέα πλευράς Μπεσέ στην αιτιολόγηση και αυτή έχει ληφθεί υπόψη, συμπεριλαμβάνεται. Αλλά ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβαστούν μόνο αν συμφωνούν τα δύο μέρη. Όχι, διαφωνώ. Χρειάζεται ένας κάποιος αυτοματισμός να ισχύει, να ισχύει έτσι ένας γενικός κανόνας που να είναι πέρα από το θέμα εξουσιοδότηση ή όχι. Διαφορετικά το σύστημα θα είναι δύσκολο στη διαχείριση του αν κάθε φορά θα πρέπει να το ζητάμε. Επίσης να υπάρξει μια προστασία των στοιχείων γενική πέρα από μια ε, ανείχνευση ειδική μεμονωμένη. Και τώρα ότι τα στοιχεία για ορισμένα στοιχεία ότι χρειάζεται και αιτολόγηση και περιορισμένη πρόσβαση για ορισμένα στοιχεία, πάνω χάρη τα εμπορικά που δεν μπορούν να δοθούν σε όλους, αυτή και αλλιώς συμπεριλαμβάνεται συμβαστική λύση. Πάμε στο άρθρο 8 τώρα. Για το ότι δεν υπερχονται μόρφωση με αυτούς τους ρυθμίσεις σε διάφορα, ε, ε, κείμενα για αγαθά που παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα για την απλοποίηση. Με την απλοποίηση τα αγαθά αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται, να μεταφέρονται. Άρα λοιπόν το άρθρο 8 θα πρέπει να διατηρηθεί. Και το είχε πει άλλωστε και η Προεδρία. Και στην τροπολογία 57 αυτό συμπεριλαμβάνεται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να προβάλλει διάφορα επιχειρήματα παρασχάρη για το λαθρεμπόριο, είτε για εμπόριο λευκής σάρκας, για θέματα ασφαλείας κλπ. Θα πρέπει να μπορεί κανείς σε παρόμοιες περιπτώσεις να ζητάει κείμενα και για έγγραφα και για πλοία που κινούνται εκτός λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα διάφορες πτυχές έχουμε που δεν αναφέρονται στις δικές μας τι τροπολογίες, ε, αλλά θα πρέπει να τα θίξουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα ήθελα να τα πω αυτά. Για να δω αυτά, αυτές οι ρυθμίσεις ε, σε ποιες χώρες ε, εφαρμόζεται. Να δούμε τις χώρες χωρίς διέξοδο στη θάλασσα. Η θέση μας είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε χώρα διαθέτει ένα λιμένα ένα θαλάσσιο λιμάνι, να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση ακόμα και οι χώρες εκείνες που έχουν τη δική του σημαία και μετά με την εσωτερική ναυσιπλοεία να ρυθμιστεί αυτό να ισχύει και η εσωτερική ναυσιπλοεία και θα πρέπει να προχωρήσει μια μελέτη επιτροπή για αυτό εδώ για την εσωτερική ναυσιπλοεία Βαντάλεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και για τις, ε, την επικοινωνία μεταξύ πληρωμάτων διαφορετικής εθνικότητας και στην εσωτερική ναυσιπλοεία χώρες ας πούμε όπως η Αυστρία που δεν έχει ακτές, που δεν έχει λιμένας, δεν ξέρω διαθέτει ε, σημαία στη θάλασσα κατάλληλη. Θα πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να συνδυαστούν και με το δίκτυο safety όλα αυτά και τότε ίσως θα πρέπει να συμμετέχει και η Αυστρία και πρέπει να μελετήσουμε την περίπτωση με το Συμβούλιο, όν όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα, να τα εγγυηθούμε με μια κατάλληλη διατύπωση. Είναι κάπως προκλητικό σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, το θέμα. Αλλά θα πρέπει την Βαντάλεν την τροπολογία για τη γλώσσα, να την, για την εσωτερική ναυσιπλοεία, να το υποστηρίξουμε. Και ακόμα για τους καπετάνιους ε, με επισκέφτηκαν, ε, θέλουν να αναφερθούν και αυτοί και ακόμα στην προσέγγιση στους λιμένες δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί έτσι η θέση μας. Χρειάζονται βέβαια ορισμένα πιστοποιητικά, στο το πούμε έτσι έκτακτα, εξαιρέσεις ε, για τους καπετάνιους εκείνους, για ειδικές κατηγορίες μάλλον καπετάνιων και χρειάζεται όμως το κατάλληλο πλαίσιο να είναι διάφανο, να μπορούμε να το ελέγξουμε άνετα κλπ. Η δικιά μου πρόταση ποια είναι. Να υποστηρίξουμε την τροπολογία Βαντάλεν που είναι μια προσθήκη στη δική μου τροπολογία 10 και έτσι μπορεί να διεξαχθεί άνετα η συζήτηση και να μην ξεχνάμε ότι μερικές φορές η παράκτεια ανασυπλοεία είναι σχεδόν εμπόδιο για την ε, ανάπλευση πλοίων γενικά και θεωρείται εμπόδιο πολλές φορές όπως λέμε. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τα πράγματα. Και εγώ αυτό που προτείνω στους αδέλφους ε, του Κοινοβουλίου να θίξουν το θέμα αυτό. Αυτά είναι τα σημεία που θα ήθελα να δούμε στις τροπολογίες. Αυτά άλλωστε προέκυψαν και από τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για μία ακόμα φορά και περιμένω τα σχόλιά σας πριν από την ψηφοφορία αύριο το πρωί νωρίς. Ευχαριστούμε κύριε Στέρξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε, ο, ο συνάδελφός μας, κύριος Ντεκράν, δεν είναι παρόν και γι' αυτό θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια την οποία έκανε να βρει ορισμένες λύσεις. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν και την έκθεση γενικά. Μερικά σημεία ακόμα πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά γενικά υποστηρίζουμε την αρχή της απλούστευσης και δει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή αυτό το περίφημο άρθρο 18 που αναφέρθηκε θα πρέπει να διατηρηθεί στη μορφή που έχει για να εδραιώσει την απλούστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για να μπορέσει να εξασφαλίσει περαιτέρω και τη νομική βάση. Άρα λοιπόν ουσιαστικά συμφωνούμε με την πρόταση. Όσον αφορά τώρα το γλωσσικό, τη γλωσσική πτυχή, είναι ένα καυτό θέμα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μέσα του συμβουλίου, στα πλαίσια του Συμβουλίου να βρούμε μια συμβαστική λύση και δεν θα ήθελα τώρα να περιοριστούμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε μία μόνο γλώσσα ή σε μία μονόπλευρη λύση δεδομένου ότι ο συνάδελφος Βαντάν αναφέρει τα αγγλικά ως γλώσσα, δεν νομίζω ότι μία γλώσσα μόνο και μία μονομερής προσέγγιση είναι η καλύτερη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να καταλήξουμε σε μια μονοπλευρη λυση δεδομενου οτι ο συναλφος βανταν αναφερει τα αγγλικα ως γλωσσα δεν νομιζω οτι μια γλωσσα μείγμα μεταξύ μιας γενικά αναγνωρισμένης γλώσσας, δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε, και μιας άλλης γλώσσας η οποία ε, θα διασφαλίζει τουλάχιστον την ασφάλεια της ερμηνείας, ας πούμε ισπανικά ή γαλλικά. Κάποια, κάποια, κάποιο μεσόωρο, κάποια συμβιβαστική λύση να βρούμε. Ο συνάδελφος κύριος Μαρινέσκο θα παρουσιάσει και αυτό στις παρατηρήσεις του όσον αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα, συμφωνούμε απολύτως με τον εισηγητή και παντού όπου αναφέρεται η ημερομηνία 2015 από πλευράς ΕΛΚ θα προτείνουμε να αλλάξει και να παραμείνει στο 2013. Ελπίζω αύριο να καταλήξουμε σε μια καλή λύση όσον αφορά την διαβίβαση ηλεκτρονικών, στοιχείων δεδομένων με ηλεκτρονική μορφή, συμφωνούμε με την πρόταση. Επιθυμούμε την απαλλαγή από την υποχρεωτική χρήση πιλότων, σκαφών πιλότων και πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουμε μία διαφανή μέθοδο που θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητές της και για να μπορέσει να έχει την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει το σύστημα της πλοήγησης με πιλότο ή όχι. Αλλά πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια έτσι ώστε να μπορούν και άλλες χώρες, άλλες πλευρές να απαλλαγούν από αυτήν την υποχρεωτική ενέργεια Πιστεύω θα καταλήξουμε λοιπόν σε ένα συμβιβασμό και σε μια ενιαία εφαρμογή, εφαρμοστική ερμηνεία. Ο κύριος Φαντρόη από την πλευρά των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μας Γκουίντο είναι, έχει κολλήσει σε ένα αεροδρόμιο στην Ιταλία και δεν είναι εδώ δυστυχώς. Καταρχάς μια γενική παρατήρηση. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή γενικά. Όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας, στο άρθρο 5 σας υποστηρίζω σε αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε προς μια ομοιομορφία και για να υποστηρίξουμε την τροποποίηση του κυρίου Βαντάλε, ο οποίος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, το, να μελετήσει αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απλώς πρέπει να μελετηθούν τα υπέρ και τα κατά. Επίσης να εξετιστούν ορισμένες ιδιαιτερότητες μπορεί να φαίνονται λίγο, λίγο παράξενες. Ε, δηλαδή να έχουμε Γερμανούς ε, καπετάνιους να μιλάνε μεταξύ του υποχρεωτικά στα αγγλικά. Ε, εν πάση περιπτώσει, η κατεύθυνση είναι σωστή. Οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν. Όσον αφορά τη θέση ενισχύ, συμφωνούμε με τον εισηγητή 2013. Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη χρονολογία και πρέπει να επιβεβαιωθεί και θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο. Μια τρίτη παρατήρηση που ανέφερε ο κύριος Γκος είναι η τροπολογία 10 που ζητεί ε, ένα ε, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πιστοποιητικά εξέξεις. Δεδομένου και πιστεύω ότι η ομάδα μου μπορεί να συμφωνήσει, δεδομένου ότι θα πρέπει, εφόσον, εφόσον ακολουθούν κοινέ διαδικασίες με αυτή την προϋπόθεση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία μέθοδο η οποία να έχει ομοιόμορφη ισχύ σε όλους. Βεβαίως αναγνωρίζουμε ιδιαιτερότητες, παραδείγματο χάρη λιμάνια, όπου είναι πολύ πιο δύσκολη η είσοδος και η έξοδος. Και πολλές φορές μπορεί οι συνθήκες να διαφέρουν ανάλογα με την παλήρια, με την άμποτη και παλήρια, ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες. Εάν λοιπόν το λάβουμε υπόψη μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Τέταρτον, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για το ότι έλεγα υπόψη την τροπολογία του κυρίου Μπάνα. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτήν. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Για τους πράσινους ο κύριος Δαφέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση Στέρξ μου φαίνεται αποδεκτή, τη δέχομαι. Είμαστε υπέρ. Εφόσον μάλιστα καθορίζει εδώ μια πραγματική απλοποίηση των δικασιών και άρα ενθαρρύνει έτσι τις θαλάσσιες μεταφορές. Και γι' αυτό ενθαρρύνουμε και εμείς τον κύριο Στέρξ να επιμείνει στην ημερομηνία του 2013 και οι δύο συμβιβαστικές προτάσεις που κάνει για την προστασία των δεδομένων και αυτές μας φαίνονται αποδεκτές. Τροπολογίες 22, 55, 56, 8, 30, 33 και 35 δηλαδή. Γενικά συμφωνούμε λοιπόν με μία μόνο διαφωνιούλα έναν περιορισμό. Όχι επί της ουσίας, αλλά aller που αφορά τη γλώσσα, διότι η διοικητική απλοποίηση δεν θα σήμαινε τίποτε αν δεν υπήρχε και μία κοινή συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων και των εταιριών και άρα η κοινή γλώσσα που προτείνεται εδώ ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αντιρρήσεις <coughs> και γι' αυτό προτείνουμε μία τροπολογία, την 9 στο σημείο 5, δηλαδή μία περίοδο μεταβατική ώστε να μπορούν και οι μικροί λιμένες με το όριο του 10% του διεθνούς εμπορίου της διεθνούς κίνησης να μπορούν να έχουν το χρόνο να δύο-τρία χρόνια για να μάθουν οι υπάλληλοι του την κοινή αυτή γλώσσα για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις και να γίνει και πιο εύκολα αποδεκτή η κοινή αυτή γλώσσα να προλάβουν δε όλοι και να τη μάθουν. Να, αυτή είναι μια αποσαφήνιση το προτείνουμε στο συμβιβασμό με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, αυτό το θέμα της γλώσσας, τη μεταβατική αυτή περίοδο λοιπόν. Κατά τα άλλα έχουμε γενικό συμφωνήσει με τον κύριο Στέρξ. Ευχαριστούμε η κυρία Φώστα για τους συντηρητικούς. Εγώ θα είμαι σύντομη. Τα έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Στέρξ. Τον ευχαριστώ εξ ονόματος της ομάδας μου για τη συνεργασία που είχαμε και για τις συναντήσεις μας. Ένα-δυο θέματα μόνο. Πρώτον, για τα σχόλια του κυρίου Μαρινέσκου για τα πολεμικά πλοία. Αυτό που είπε γενικά το υποστηρίζουμε, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω να εμφαίνεται σε κανονισμό η οδηγία γιατί τα στρατιωτικά θέματα εξαιρούνται εξορισμό. Όσο για τη χρήση της Αγγλικής, συμφωνώ με τον κύριο Στέρξ, το θέμα είναι πώς θα υπάρξει λιγότερη δυνατή σύγχυση και μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Και αυτό σκοπεύει νομίζω η χρήση της Αγγλικής. Βέβαια, Υπάρχουν πολλή γλώσσα πληρώματα, αλλά οι περισσότεροι ήδη μιλάνε αγγλικά. Λοιπόν, εκεί που διαφωνούμε όμως είναι η ημερομηνία θέσεως ενισχύει. Εμείς θα θέλαμε το 15 για να μπορέσουν όλες οι χώρες να, έχουν, να προετοιμάσουν τον καινούριο τους προϋπολογισμό για να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις. Γενικά όμως παρά τις δύο αυτές παρατηρήσεις που είχα να κάνω, νομίζω ότι αύριο κατά την ψηφοφορία θα στηρίξουμε γενικά την έκθεση. Ευχαριστώ. με, ο Αντιπρόεδρος Ρίκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρτήρια στον κύριο Στέρξ ε, για την άριστη αυτή έκθεση σε τόσο περίπλοκο θέμα. Ορισμένε παρατηρήσεις ε, και μια αλλαγή στις ε, τροπολογίες μου. Το λεπτότερο θέμα που είναι το θέμα της γλώσσα. Διαφορά υπήρχε, υπάρχει ανάμεσα στην κοινή γλώσσα και στη γλώσσα αναφοράς. Χρειάζεται μια γλώσσα αναφοράς για τους λόγου που ακούσαμε, αλλά άλλο είναι όμω η κοινή γλώσσα Βέβαια, ορισμένε φορέ θα έχουμε και μια κάποια ανταλλαγή και από, γερμανικά σε γερμανικά, από ολλανδικά σε ολλανδικά, γιατί να μιλάνε μια άλλη γλώσσα, μια τρίτη γλώσσα. Δεν χρειάζεται. Και το πνεύμα τη όλης οδηγίας ποιο είναι. Αυτά τα πράγματα να απλοποιηθούν πρώτα για μια επιπλέον υποχρέωση η οποία ε, θα, ίσχυε, και τώρα ε, θα ήθελα να είναι τώρα θεσμικό το θέμα με, με τη γαλλική γλώσσα επειδή δεν πάει με το Σύνταγμα και θα προδημούσε ένα κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη σύγκληση και τη συμφωνία με τον εισηγητήριο πάντων. Γι' αυτό την τροπολογία 38 θα ήθελα να διαγραφεί, αλλά η 50 μου να διατηρηθεί, γιατί ο συντονιστή μα όπω ε, περιέγραψε, εδώ έτσι μπορούμε να τα ζητήσουμε ισορροπημένα με το Συμβούλιο και το ίδιο είπε άλλωστε και ο εισηγητής για να ανοίξουμε δρόμο για το μέλλον και δεν είναι κάτι το απομονωμένο από τη μία την άλλη πλευρά. Κάτι ακόμα. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητού και η τροπολογία 48 να διαγραφεί η όλη συζήτηση που διεξήχθη με τη Συμβούλιο και την Επιτροπή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Συμφωνούμε με αυτό λοιπόν και η πρόταση αυτή είναι καλύτερη ακόμα και από την τροπολογία μας. Και επίσης να διαγραφεί 40 για, την, για το χειρισμό των πλοίων και ακόμα δύο πραγματάκια αν γίνεται αυτό ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη στην τροπολογία 30 μετά από την ημερομηνία 2013 να διατηρηθεί για τη συνέχιση διατήρηση μεταβίβαση από το στοιχείο μετά το 2013 να ψηφίσουμε ξεχωριστά το πρώτο μέρος από το δεύτερο μέρος λοιπόν της τροπολογίας αυτή. Και συμμερίζουμε αυτό που λέει η για την ημερομηνία όλοι και εκτός από τον εισηγητή θα ήθελαν η εφαρμογή να γίνει όσο γίνεται ταχύτερα. Αλλά πλευρά τακτική τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να ξεκινήσουμε με μια μαξιμαλιστική θέση απέναντι στο Συμβούλιο και να πούμε το 2013, γιατί ξέρουμε το Συμβούλιο υποστηρίζει, έχει σαν βάση του την ημερομηνία τη χρονιά 2017. Αλλά λοιπόν εντάξει να πάμε μετά στο 2015 η πρόταση αυτή είναι πιο ρεαλιστική σε σχέση με το Συμβούλιο. Όπω δεν πήγε Φούστερ, λαμβάνει υπόψη τη και το τι υποχρεώσει υπάρχουν και τι προβλήματα από τεχνική πλευρά για την εφαρμογή αυτού του συστήματο, για την κατάστασή του, όπω έχουν σήμερα τα πράγματα και η κατάσταση. Και τι γίνεται τώρα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρή η θέση μα από το ξεκίνημα ήδη και μετά σιγά σιγά να πούμε εντάξει δύο χρόνια παραπάνω είτε να πούμε από την αρχή 2015. Θέμα τακτικής λοιπόν να το συζητήσουμε. Thank you. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος κ. Φαντάλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να ευχαριστήσω την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα ιδίως ε, επί της τροπολογίας ε, για τις εξαιρέσεις. Υποστηρίζω την ε, πρόταση σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να ρωτήσω το ΕΛΚ να ξανακοιτάξει τις τροπολογίες μου για τη χρήση της γλώσσας. Τις έχω διατυπώσει πολύ προσεκτικά για να μπορέσει η Κομισιόν επίσης να τις μελετήσει Καταλαβαίνω την ε, παρατήρηση του συναδέλφου αν θα πρέπει τελικά δύο Γερμανοί καπετάνοι να επικοινωνούν στα αγγλικά. Αλλά έχω υποβάλει αυτές τις τροπολογίες επί έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα και δεί μοιραία ε, επειδή υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να δράσουν έγκαιρα και άμεσα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και κάνω μια έκκληση στον, και στον εισηγητή και στο ΕΛΚ να ξαναμελετήσει τις τροπολογίες μου για τη γλώσσα. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν δύο πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες που έχω υποβάλει. Στη σύμβαση ορίζεται το εξής. άφηξη και αποχώρηση πλοίων. Αυτά τα δύο, οι δύο ενέργειες, οι δύο δραστηριότητες, άφηξη και αποχώρηση είσοδος και έξοδος. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα λάβουμε υπόψη και θα καλύψουμε και τη διαμονή, τον ελιμενισμό του πλοίου και θα λέει arrival, stay and departure, δηλαδή άφηξη, ελιμενισμός, διαμονή και αποχώρηση, έξοδος. Αν θα καλύψουμε δηλαδή και την τρίτη πτυχή. Η ίδια σύμβαση πολύ συγκεκριμένα αποκλείει τα πολεμικά πλοία, ενώ η οδηγία αναφέρει τον ορισμό του πλοίου ως ε, όχι, πλοίο το, πάσης μορφής. Ε, ε μέσο μεταφοράς πάσης μορφής. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ότι ε, θα, ήθελα να ζητήσω συγκεκριμένα να αποκλειστούν τα πολεμικά πλοία από αυτή την οδηγία. Ο κύριος Καλομίτσος από την Κομισιόν. Thank you, thank Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ δε ιδιαίτερα τον εισηγητή για την συνεπέστατη αυτή ανάλυση. Ξέρουμε ότι είναι ο κύριος εμπειρογνώμονα σας για αυτά τα θέματα και η έκθεσή του είναι λογικότατη. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, δύο-τρία είναι τα κύρια προβλήματα. Πρώτον, η ημερομηνία. Γιατί είπαμε το 13 και γιατί επιμένουμε ότι είναι λογικότερο το 13 και διαφωνούμε απόλυτα με το Συμβούλιο. Διότι υπάρχουν δύο τεχνικά θέματα εδώ, δύο οδηγίες, δύο νομικά κείμενα ας πω, που πρέπει να εφαρμόσουν, όπου, σύμφωνα με τα οποία πρέπει τα κράτη να εφαρμόσουν όλες τις τεχνολογικές αλλαγές με διαμιάς. Η μία, το ένα από αυτά είναι η οδηγία για τις θαλάσσιες μεταφορές και το άλλο η οδηγία που αφορά το σύστημα ασφαλείας, το δίκτυο ασφαλείας στα πλοία. Πρέπει τα πλοία να δίνουν ανα πάσα στιγμή το στίγμα τους κτλ. Έχουμε λοιπόν 713-714 σταθμούς στην Ευρώπη που παίρνουν αυτές τις πληροφορίες και με το κέντρο ΕΨΑ στη Λισαβόνη και τα δύο περιφερειακά κέντρα, το ένα στη Βαλτική κοντά στην Κοπεχάγη και το άλλο κάπου αλλού, έχουμε ήδη πολύ καλό σύστημα επιτήρησης για να παίρνουμε το στίγμα των πλοίων και το 2013 υπάρχει υποχρέωση, προβλέπεται, να αρχίζει να εφαρμόζεται το σύστημα ΙΤΑ δασμών. Δηλαδή, οι πληροφορίες για τα αγαθά που μεταφέρονται, για τα επικίνδυνα αγαθά, αυτά καλύπτονται ήδη από την άλλη οδηγία και άρα τεχνικά ήδη υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να έχουν εφαρμόσει, καταστήσει τις υποδομές για αυτές τις δύο οδηγίες. Αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω λόγος για παραπάνω επενδύσεις εκτός από διοικητικέ. Άρα δεν παρεμποδίζεται η εφαρμογή το 2013. Στο Συμβούλιο χάσαμε. Αλλά θέλουμε τώρα να μας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, να γίνει νωρίτερα η εφαρμογή, αλλιώς δεν είναι λογικό να απλοποιούμε τα πράγματα αλλά μετά να καθυστερούμε. Δεύτερο πρόβλημα, τα λιμάνια, το, η γλώσσα μάλλον στα λιμάνια. Και εδώ θα προσπαθήσω να μην περιοριστώ μόνο στο τεχνικό μέρος. Το Συμβούλιο έχει πει ότι τουλάχιστον όχι προφορικά αλλά τα δεδομένα που θα υποβάλλονται γραπτός γιατί έτσι κυρίως θα μεταφέρονται τα δεδομένα, γραπτός δηλαδή μεταξύ πλοίου και ακτής, να είναι στην κοινή γλώσσα που ήδη χρησιμοποιούν όλοι, η αγγλική δηλαδή, στην αγγλική. Πράγματι η κοινή γλώσσα <coughs> για λόγους επικοινωνίας είναι η αγγλική, αλλά για προφορική επικοινωνία νομίζω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες. Εξήγησε ο εισηγητής τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Θα σήμαινε ρωσικά και δύο-τρεις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρέως στις θαλάσσιες μεταφορές, γιατί χρησιμοποιούνται μόνο τα αγγλικά, καμιά φορά και τα γαλλικά και το Σόλας ήδη έχει πει ότι τα αγγλικά πρέπει να είναι και η γλώσσα επικοινωνίας εκτός από τις γραπτής υποβολής δεδομένων. Αλλά αυτό γιατί εκείνοι ήδη κάνουν και εκπαίδευση στα αγγλικά. Και θα υποχρεώνονταν έτσι οι υπάλληλοι των λιμένων να κάνουν μια τουλάχιστον βασική εκπαίδευση στα αγγλικά. Ξέρετε ότι πολλές φορές στα πληρώματα δεν υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας και είναι πρόβλημα αυτό οι περισσότεροι δε επιλέγουν τα αγγλικά. Γι' αυτό υποχρεώνουμε μία κάποια ελάχιστη γνώση τους, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι υπάρχουν δύο διεθνείς συμβάσεις που ήδη μιλούν για την κοινή γλώσσα της ναυτιλίας να πείτε; Τώρα, τα πιστοποιητικά. Ε, οι εξαιρέσεις μάλλον από τα πιστοποιητικά του καπετάνιου του παίλοτ μάλλον. Το είχαμε προτείνει ήδη δυο φορές αλλά δεν είχε εγκριθεί. Τώρα αν ο εισηγητής και το κοινοβούλιο το δέχονται γιατί όχι, αν δεν το έχουμε βάλει μέσα στο κείμενο, στο κύριο σώμα της οδηγίας, αλλά είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τέλος, ο κατάπλους και απόπλους και η παραμονή του πλοίου στο λιμάνι στη σύμβαση, σε προηγούμενες συμβάσεις αναφέρεται επίσης η διαμονή αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Μερικά πλοία μπορούν να μένουν πάρα πολύ καιρό στην Αφρική πριν αποπλέψουν αλλά συνήθως στην Ευρώπη η παραμονή στο λιμένα είναι πολύ μικρή. Τέλος πάντων, ίσως είναι κάτι που δεν χρειάζεται, αλλά απ' την άλλη δεν θα έχουμε και καμία στεναρή αντίρρηση. Τέλος τα πολεμικά. Τα πολεμικά αποκλείονται ρητά από την οδηγία αυτή και για την παρακολούθηση και για τα στίγματα και για όλα αυτά αποκλείονται. Εξορισμού εμείς δεν καλύπτουμε σε τέτοιες οδηγίες και τα πολεμικά διότι αυτά τα αφορούν άλλα νομοθετικά κείμενα της Ένωσης. Αν όμως επιμένετε και λέει, θεωρείτε ότι αυτό θα αποσαφήνιζε τα πράγματα περισσότερο, δεν νομίζω θα υπήρχε καμία ιδιαίτερη δυσκολία και γι' αυτό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κρατήστε το 2013 και μην αρχίσετε με το 2015 γιατί τελικά θα καταλήξουμε στο 16-17. Αρχίστε με το 2013. να για να καταλήξουμε ίσως στο 15. Για τη γλώσσα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία. Στην πράξη όμως πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν όλοι με κάποια κοινή γλώσσα, όπως γίνεται και στην αεροπορία, δηλαδή στα αγγαλικά και για τα πιστοποιητικά εξαιρέσεων των πιλότων, των pilots, και αυτό νομίζω είναι εύκολο να λυθεί. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτε. Αν ξέχασα με συγχωρείτε. Ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα ερωτήματα που τέθηκαν προς την Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Μήπως κύριε Στέρξ θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να κάνω μία-δύο παρατηρήσεις για όσα είπε ο συνάδελφος Ελκαντράουι. Ναι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τεράστιες τοπικές διαφορές. Και μετά οι τοπικές αρχές οι οποίες εκδίδουν το πιστοποιητικό αυτό ακολουθούν σειρά ολόκληρη ρυθμίσεων που ισχύουν. Και πολλοί από τον κόσμο αυτό διαμαρτύρονται, παραπονιούνται για τα πιστοποιητικά αυτά, γιατί έγιναν λάθη και δεν έγιναν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, με αποτεσματικό τρόπο. Ε, θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερα την παράκτια αυτοπλοεία και για την ημερομηνία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το 2013 ή να απομακρυνθούμε όσο γίνεται λιγότερο αναφέρθηκε το θέμα των τελωνίων, το ένα το άλλο. Εμείς όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο γίνεται ταχύτερα να απλοποιήσουμε και ελπίζω να με υποστηρίξετε. Για να δούμε και με τη γλώσσα τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε ποια είναι η σύστασή μου. Ξέρω επίσης ότι είναι δύσκολο το θέμα αλλά αυτό όπως είπε ο κ. Βαντάλ είναι πολύ σημαντικό στην αυσιπλοεία υπάρχουν σήματα ε, και θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε και με το Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε, εντάξει, ίσως το κείμενο το οποίο αύριο θα ψηφίσουμε, ε, ίσως να μπορέσω να σας το υποβάλω και για τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, αλλά ε, εδώ με τη Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλύει ψηφοφορία θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και πάλι. Ελπίζω να τύχω τις υποστηρίξεις σας για το επόμενο, για το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί 9 και 10 θα ψηφίσουμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ναυτιλιακή πολιτική και η στρατηγική στόχη μέχρι το 2018 εξέταση τροπολογιών. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σ' αρχίσω με, ευχαριστώντας καταρχάς όλους μου τους συναδέλφους, 99 τροπολογίες έχουμε. Χαίρομαι, γιατί αυτό δείχνει ακριβώς τη σημασία αυτού του θέματος, με το οποίο ασχολούνται όλοι ενδελεχώς. Την τελευταία φορά Είχα ομαδοποιήσει τις τροπολογίες γύρω από τα βασικά σημεία μαζί με τον σκιώδη εισηγητή για να παρουσιάσουμε την ε, τελική, τον τελικό κατάλογο ε, τροπολογιών για την ψηφοφορία. Τα βασικά θέματα, πρόεδρε, είναι τα εξής. Και θα τα δείτε στις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ελπίζω να τις έχετε. Καταρχάς, τη διασύνδεση μεταξύ ναυτιλιακών κομβικών σημείων και των δημοσιονομικών αναγκών που χρειάζονται. Και πιστεύω ότι το εδάφιο Α το καλύπτει. Ε, να δούμε λοιπόν ακριβώς πώς θα εξασφαλίσουμε την διασύνδεση και τις υποδομές μεταξύ των λιμένων και των, το, του εσωτερικού της χώρας και των λιμένων. Υπάρχουν και πολλές άλλες τροπολογίες τις οποίες δεν έχω συζητήσει με όλους. Απλώς θα παρουσιάσω τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Σας είπα ότι αυτός ήταν ε, η συμβιβαστική τροπολογία Α, η Β, Voor gelden, belangstelling Όπου εστιάζουμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στο πώς θα προσελκύσουμε νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι μαζί με συναδέλφους έχουμε διατυπώσει ένα καλό κείμενο στο συμβιβασμό Β και καλύπτουμε πολλές, ε, πολλά αιτήματα συναδέλφων. Το ίδιο ισχύει και για τη συμβαστική τροπολογία Γ. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες με παρόμοιες διατυπώσεις όσον αφορά τη σύμβαση του ILO και την εφαρμογή της του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και πολλές τροπολογίες βεβαίως παρουσιάζουν διαφορετικές, διαφορετικά αιτήματα. Το συμβιβαστικό κείμενο Γ πιστεύω τώρα ότι καλύπτει επιτυχώς δύο-τρεις πολιτικές ομάδες. Εν συνεχεία, συμβιβαστική τροπολογία Δ. Ξέρω ότι εδώ υπάρχουν ακόμα διαφορές απόψεων. Θα προτιμούσα το δικό μου κείμενο, προφανώς. Διότι πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα bonus Άλλοι λένε ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε να υιοθετήσουμε μια τέτοια ιδέα. Προς όφελος λοιπόν του συμβιβασμού είπα ότι θα δεχτώ τη συμβιβαστική τροπολογία παρόλο που πιστεύω ότι η δική μου διατύπωση είναι καλύτερη. Στην συμβιβαστική τροπολογία Δέλτα λοιπόν θα δείτε ότι στον κατάλογο ψηφοφορίας λέω ότι προτιμώ το δικό μου κείμενο και γι' αυτό προτείνω ξεχωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα δείτε όταν παλάβετε τον τελικό κατάλογο ψηφοφορίας. Το split vote που ζητώ. Θα εξηγήσω λοιπόν τη θέση μου όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. Να δούμε πώς θα πάει λοιπόν τώρα η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά την πειρατεία, την πειρατεία. Εδώ και πάλι πολλοί συνάδελφοι, χωρίς να το συζητήσουν μεταξύ τους, έχουν υποβάλει τροπολογίες που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Και θέλουμε να διευκρινίσουμε τη θέση μας επί της πειρατείας και να αναφερθούμε στην επιτυχή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον αυτής της πειρατείας. Υπάρχουν 5-6 τροπολογίες που, είναι πάρα, που μοιάζουν πάρα πολύ. Και αυτό το πρόσεξα μόλις τις ε, διάβασα και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να δεχθούμε τον συμβιβασμό ε, τη συμβιβαστική τροπολογία ε. Εν συνεχεία υπάρχουν και άλλες τροπολογίες πρόεδρε Ένας συνάδελφός μας, ο κύριος Τούσας, έχει υποβάλει σειρά τροπολογιών που βρίσκει δεν είναι εύκολο να τις υποστηρίξω, διότι πιστεύω αποκλίνουν από το στόχο μας που είναι η κοινή πολιτική. Έχω μία διαφορετική άποψη, ζητώ συγγνώμη λοιπόν έναντι του συντάκτη των τροπολογιών αυτών και αυτό θα το δείτε στον κατάλογο των, ε, της ψηφοφορίας των τροπολογιών. Εν συνεχεία, ο κύριος Μπασέ έχει μία σειρά τροπολογιών. Ας δούμε την 54. Στην 54 την συζήτησα με αρκετούς συναδέλφους την τελευταία εβδομάδα, τροπολογία 54 Μπασέ, και είναι ένα σύστημα εμπορία εκπομπών τη ναυτιλία, το οποίο θα λειτουργεί ω συμπληρωματικό εργαλείο στον κατάλληλο τη ψηφοφορία, Μα έχω βάλει συν ή πλην. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα αυτό που πρέπει να εξετάσει η Κομισιόν. Και ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, το επεξεργάζονται αυτό το σύστημα, έχει ξεκινήσει, έχουν κάτι συγκεκριμένο για αυτό το σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να, να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Καραμίτσου για αυτό το συγκεκριμένο θέμα που καλύπτει η τροπολογία 54, παράγραφος 13α, νέα. Και έτσι θα μπορέσω και εγώ να διαμορφώσω την τελική μου άποψη για την ψηφοφορία. Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν έχω καλύψει τα πάντα. Υπήρξε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας. Έχουν, έχουμε σε πάρα πολλά σημεία συγκεράσει τις απόψεις μας, έχουμε επιτύχει συμβιβασμούς και το απόγευμα θα λάβετε την τελευταία μου πρόταση για να είμαστε έτοιμοι στην ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον εισηγητή. Ο κ. Κουμουτσάκος από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ε, η στρατηγική για την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Θαλασσίων Μεταφορών για το 2018 είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Ειδικά στην παρούσα διεθνή αρνητική συγκυρία ενώ οικονομική ε, αρνητική συγκυρία. Ο Σάλφος κ. Βαντάλεν έκανε μια πολύ καλή δουλειά με πραγματική διάθεση για συνεργασία και αναζήτηση σύνθεσης απόψεων. Και ε, τον ευχαριστώ για την ε, επικοδομητική του αυτή στάση. Έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ένα πολύ ισορροπημένο και θετικό κείμενο Τέσσερα βασικά επιμέρους ζητήματα απασχόλησαν αυτό το, απασχολούν αυτή την έκθεση. Πρώτο, η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Νομίζω ότι το κείμενο καλύπτει επαρκώς αυτή την σοβαρή ανάγκη, ειδικά σε μια περίοδο που τρίτες ε, χώρες πολλές φορές καταφεύγουν σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό και γι' αυτό η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας πρέπει να υποστηριχθεί. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να υποστηριχθεί και το μέτρο των κρατικών ενισχύσεων, state aid. Και αυτό το καλύπτει ε, επαρκώς η έκθεση Βαντάλερ. Το δεύτερο ζήτημα είναι το πρόβλημα κάλυψης των αναγκών σε ψυχοδυναμικό δυναμικό της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Και βεβαίως η ανάγκη προσέλκυσης καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και υψηλού επίπεδου προσωπικού. Ως προς αυτό ε, έχουμε παρουσιάσει ε, και ε, έχει παρουσιάσει και ο Μιλών αλλά και άλλοι συνάδελφοι από το ΕΠΠ συγκεκριμένες τροπολογίες οι οποίες βλέπω ότι αντιμετωπίζονται θετικά από τον εισηγητή. Το τρίτο ζήτημα είναι η συμβολή των θαλασσίων μεταφορών στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής αν και το τμήμα επιβάρυνσης που αναλογεί στις θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ μικρό, είναι βέβαιο ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς όμως, και το τονίζω αυτό, να πλήττεται με τρόπο αντιπαραγωγικό και πέραν του λογικού η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας που παραμένει και το πρώτο και μεγάλο ζητούμενο. Ε, επίσης εκεί θεωρώ ότι έχουμε ε, καταφέρει να έχουμε μια συναντήληψη στην πλειοψηφία και ε, το κείμενο και οι προταθήσεις τροπολογίες να μην παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τέλος, το θέμα της πειρατείας. Ε, ζητήσαμε από πολύ νωρίς να είναι το κείμενο της, ε, της έκθεσης πιο φιλόδοξο από ό,τι ήταν το αρχικό κείμενο που παρουσίασε ο εισηγητής, ο, ο ραπορτέρ. Νομίζω και εκεί ότι έχουμε πετύχει μια καλή ισορροπία. Σε όλους αυτούς τους τομείς και στους τέσσερις που ανέφερα, τόσο ο Μιλών όσο και οι άλλοι συνάδελφοι από το ΕΠΠ έχουν καταθέσει ουσιαστικές και σοβαρές τροπολογίες που βοηθάνε να πάει το συνολικό κείμενο προς σωστή κατεύθυνση. Ε, δεν έχω κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις για να σας πάρω περισσότερο το χρόνο. Νομίζω ότι οδεύουμε προς μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τους σοσιαλιστές ο κύριος Φλάνκενστάιν. Πρόεδρε, κύριε Βαντάλεν, αγαπητοί συνάδελφοι, και εμείς ευχαριστούμε τις εργασίες όλων αυτών που συνέβαλαν στην υποβολή 99 τροπολογιών. Γενικά έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο που μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο, όμως έχουμε ακόμα μερικά θεματάκια τα οποία εκκρεμούν. Πρώτον, κύριε Βαντάλεν, εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε κατά τη γνώμη σας, ε, προς τα πού κλείνετε στη συμβιβαστική τροπολογία Β. Ε, λέτε ότι είναι πιο καλύτερη ο συμβιβασμός ε, Β έναντι της τροπολογίας 22 για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, τον κύριο Μπεσέ, θα θέλαμε να ξέρουμε σχετικά με την τροπολογία 24 πώς τι ακριβώς εννοεί διότι κατά την άποψή μας αυτές οι conferences όπως λέμε στις θαλάσσιες μεταφορές ε, δεν υπάρχουν πια ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί που λέει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θαλασσίων μεταφορών. Εν συνεχεία Περιμένουμε πάρα πολύ με ανυπομονησία και ενδιαφέρον την ε, πρόταση της Κομισιόν για την, ε, το συμψηφισμό, την ανταλλαγή ε, εκροών και εκπομπών Και τέλος είπατε ότι δική σας, ε, το δικό σας αρχικό κείμενο όσον αφορά την, το συμβιβασμό ε, προτιμάτε το αρχικό σας κείμενο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου, πείτε ακριβώς πού, σε ποιο σημείο προτιμάτε τη δική σας διατύπωση. Και στον συμβιβασμό σας ε λατινικά, σίγμα ταφ ελληνικά, πιστεύουμε ότι πρέπει να προσθέσουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 82, διότι δεν υπάρχουν μόνο ε, πολιτικές και στρατιωτικές πτυχές, αλλά ε, στο μέλλον μπορεί να επισέλθουν και κοινωνικά, κοινωνικοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες και θα πρέπει να περιληφθούν και αυτές οι κοινωνικοπολιτικές πλευρές. Είπατε ότι θα υποβάλλετε μία προφορική τροπολογία από τις τροπολογίες 99 γιατί πιστεύετε ότι ένα λεπτό να που είμαστε Πιστεύετε ότι θα συνεργαστείτε καλά με την Επιτροπή Ναυσιπλοείας του Ρήνου, επειδή αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία, και θα ήθελα να σας θυμίσω, δεν υπάρχει μόνο ο Ρήνος για την εσωτερική ναυσιπλοεία, αλλά και ο Δούναβης, ο Έλβας και άλλα ποτάμια. Να το προσέξετε αυτό, μήπως τυχόν και δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Το ΕΛΚ μας παρακάλεσε να αλλάξουμε την τροπολογία μας 26, που αφορά, αφορά τα κοινωνικά πρότυπα πρότυπα σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις. Καλύτερα να πούμε promoting λοιπόν. Προωθεί, προωθεί. Πρέπει να αντί προωθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Φλέγκεστάιν. Η κυρία Μάισεν από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Σάβησα, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια, είναι καθοδόν. Έρχεται και δεν μπορεί να μιλήσει ίδια. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Βαντάλεν, για την πολύ φιλόδοξη έξεση του. Ε, σας γνωρίζουμε ότι είσαστε άνθρωπος της θάλασσας, άνθρωπος του νερού. Και γι' αυτό λοιπόν ε, κάνατε αυτό το εξαιρετικό έργο και σας ευχαριστώ και εξ ονόματος της κυρίας Σαβισάρ που λάβατε υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Έτσι καταλήξατε σε 99 τροπολογίες. Βλέπετε ότι ως πολιτική ομάδα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνωμοδότηση και συνεργαστήκαμε θαυμάσια για την προετοιμασία. Πράγματι, εμείς την ομάδα μας προσέχουμε ιδιαίτερα την σημασία της ναυσιπλοείας. Ότι δηλαδή η ναυσιπλοεία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός τομέας και ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα της ε, ασφάλειας, δεδομένου ότι η ναυσιπλοεία παίζει έναν ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη το 41% του διεθνούς ε, στόλου είναι ευρωπαϊκός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλη τη σημασία και θέλουμε να την τονίσουμε. Ταυτόχρονα θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ε, βλαβερών αερίων, θέλουμε να ε, προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά πιστεύω ότι η τροπολογία 54 είναι πολύ περιοριστική διότι αναφέρει το έτος 2010 δεν, δεν ε, συμβαδίζει, δεν συνάδει αυτή η χρονολογία με άλλες ε, οριζόντιες ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε υιοθετήσει. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουμε το 2010 στην τροπολογία 54. Βέβαια θέλουμε καθαρή ναυσιπλοεία, καθαρά λιμάνια, αυτό είναι σαφές. Επίσης, χρειαζόμαστε μια εξαιρετική κατάρτιση, μια ναυτιλιακή εκπαίδευση, η οποία να καλύπτει τις μελλοντικέ μας ανάγκες. Αυτό καλύπτεται θαυμάσια από την ε, πρότασή σας. Όσον αφορά την πειρατεία, πιστεύω ότι έχετε καλύψει το θέμα αυτό ε, ε, ευρέως στην έκθεσή σας, δεδομένου ότι αναφέρεστε ότι πολλοί στόλοι έχουν πρόβλημα με την πειρατεία. Όσον αφορά το Ρήνο, μετά την παρατήρηση του κυρίου Φλέκενστάιν, εγώ μένω πιο κοντά στον ποταμό Ελβά από ότι στο Ρήνο. Εν πάση περιπτώσει, αναξάρτητα από ποιο ποτάμι ε, συζητούμε, καλύτερα είναι να έχουμε τώρα μία έξεση η οποία να αναπτύξει την ε, ναυσιπλοεία μέχρι το 2018 χωρίς να αναφέρει στο θέμα της εσωτερικής ναυσιπλοείας συγκεκριμένα ποτάμια. Γενικά λοιπόν να το αφήσουμε. Ε, εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ εμπεριστατωμένη και εξαιρετική έκθεση και πιστεύω ότι θα υπερψηφιστεί αύριο και θα δείχνει και την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε γενικά στον τομέα των μεταφορών και ειδικά στην αυσιπλοεία, στην αυτιλία. Ο κ. Μπεσέ, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες επιφυλάξεις για την έκθεση του κ. Βεντέλ. Θα τον υποστηρίξουμε με την ψήφο μας αύριο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η σημαντική λύση του κ. Βαντάλεν για θέματα πειρατείας. Μας αρέσει. Δύο σημεία όμως θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε στα πλαίσια της συζήτησης που έχουν να κάνουν περισσότερο με την Επιτροπή παρά τον εισηγητή. είναι η αγορά εκπομπών. Θα πρέπει να δούμε τι θα ήθελα να κάνει γι' αυτό η Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος τι φρονεί σχετικά. Σημαντικό όμω είναι στην έκθεση να εμφανιστεί και ο στόχος ότι και στην αυτιλία θα πρέπει να δίνουν εκεί τη μάχη τους ε, όπως και οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς που θα πρέπει να μπουν στην ίδια βάση όλοι δίνοντας την εξίσου τη μάχη τους και για την 54 τροπολογία εκεί αυτό αφορά και ακόμα για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα για την Επιτροπή το Μητρό το Ευρωπαϊκό από παλιά, από ό,τι μου λένε ήδη το ακούμε αυτό, δεν είναι κάτι που πρώτο εμφανίζεται. Και αυτό στην έκθεση του κ. Βαντόλεν είχαμε μια τροπολογία για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό το Ευρωπαϊκό Μητρό αποτελεί εργαλείο και μάλιστα άριστο για τις ε, σημαίες ευκαιρίες, ευκαιρίας που ο στόχος μας είναι όλων μας να καταπολεμήσουμε. Ο κ. Τούσας. Μας είχε δοθεί και την ε, τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής να τοποθετηθούμε επί του συνόλου της σχετικής πρότασης με τη θέση μας. Πανερχόμενοι καταρχήν στο σύνολο της πρότασης πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ότι κριτήριο αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας και τους συναφείς κλάδους σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των λαϊκών αναγκών, του περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα και με προεκτάσεις ακόμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ειρήνη. Και αυτό το τελευταίο έχει να κάνει με την πειρατεία και όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, παρακολουθώ τις εξελίξεις από το 1980. 25 χρόνια μετά από την πρώτη φάση της κοινή ναυτιλιακής πολιτικής διαπιστώνω ότι μονότονα επαναλαμβάνεται το εξής γεγονός. Ζητήματα που κατά κόρο έχουν βάλει οι εργαζόμενοι και οι φορείς τους τα αφήνεται ως πλειοψηφία κομμάτων για την επόμενη περίοδο που θα επαναξαρτηριστεί η πορεία της κοινή ναυτιλιακής πολιτικής. Και εδώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει από κανέναν ότι τα χρόνια που έτρεξαν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ναυτιλίας και των συναφών κλάδων αποκόμισαν τεράστια αστρονομικά κέρδη. Ήδη ακόμα και σε φάση κρίσης κερδίζουν τεράστια ποσά. Όχι όλοι. Και είναι προφανώς ότι μεγάλες, μικρές επιχειρήσεις πλήττονται, συνθλίβονται και ορισμένε από αυτέ καταστρέφονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε τώρα στο βασικό επιχείρημα του εισηγητή που είπε ό,τι αφορά τι προτάσει μα. Είπε ο εισηγητή, οι προτάσει του κυρίου Τούσα, και προφανώ δεν είναι του κυρίου Τούσα μόνο, αλλά και άλλων συναδέλφων μέσα από την ομάδα, κινούνται σε μια άλλη συνολική λογική. Συμφωνούμε όλοι στο κύριο ότι πρέπει ως ελάχιστο να εφαρμοστεί η Διεθνή Σύμβαση του 2006 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε ό,τι αφορά τους ναυτεργάτες. Όλοι συμφωνούμε. Πώς θα γίνει όμως αυτό, εδώ καταγράφεται τόσο από την πρόταση της Επιτροπής, όσο και από τις τροπολογίες που είναι πρόταση à la carte. Δεν έχει καμία σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο και μιλάμε, προσέξτε εδώ, θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί προφανώς απευθυνόμενοι σε στελέχη. Μιλάμε για δικαιώματα της δεκαετίας του 1970. Δεν θέλετε να αναγνωρίσετε δικαιώματα του 1970. Αυτή είναι η ουσία. Δεν μιλάμε για κάτι καινούριο. Μιλάμε για μια διεθνή νομοθεσία που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1970. Και έχουν να κάνουν με τους όρους δουλειάς, με τις συνθήκες δουλειάς, την ασφάλεια των εργαζομένων, τις οργανικές συνθέσεις, το περιβάλλον και μια σειρά άλλου τομεί. Να λοιπόν ότι ο ισχυρισμό σα στην αντίκρουση των θέσεών μας είναι ανυπόστατο. Γιατί, για αποδείξτε μας ότι έχουμε μισάδικο. Τι λέμε απλά μέσα από την τροπολογία μας, τη συγκεκριμένη, την τροπολογία 43. Να σας τη διαβάσω. Τονίζει την ανάγκη να επικυρωθεί άμεσα και να εσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών η Σύμβαση Ναυτικής εργασία, που επικυρώθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ΔΟΕ, στις 23 Φλεβάρι 2006, που θέτει τα ελάχιστα όρια για την εξασφάλιση βασικών δικαιωμάτων των αφεργατών, ιδιαίτερη σημασία ζήτημα είναι η εσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες και του μέρους Β της σύμβασης που εμφανίζεται ως μη υποχρεωτικής εφαρμογής καθώς και εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης 145 περί συνεχούς απασχόλησης των αφεργατών η θέσπιση επίση όριμων ετοιμάτων του ναυτεργατικού κινήματο, όπω η αύξηση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, η θέσπιση του 7ου, 35ου κλπ. κλπ. Να μην πω λόγο. Γιατί δεν θέλετε, για πετε μα τα επιχειρήματά σα. Δεν θέλετε να υλοποιήσετε το διεθνέ δίκαιο τη δεκαετία του 1970. Νομίζω ότι και είναι ξεκάθαρο ότι μας, ε, με αφορά, γιατί δεν μπορώ να μιλάω και εξ ονόματος συνολικά της ομάδος, ότι δεν είναι ότι δεν έχετε ε, άποψη για τις προτάσεις μας, ε, για τις θέσεις μας. Φυσικά κινούνται σε μια άλλη ε, διαφορετική λογική που έχει να κάνει σχέση ότι αυτός ο στρατηγικής σημασία τομέα πρέπει να είναι επιοφελής για τη συντριβική πλειοψηφία των λαών και για την ανάπτυξη των λαών. Να είμαι πιο συγκεκριμένος τώρα. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 16 που έχει γίνει, θα ήθελα να γίνει split vote γιατί νομίζουμε ότι υπάρχει το ζήτημα της αντιμετώπισης των σημερών ευκαιρίας. Δηλαδή, στην τροπολογία 16 να γίνει το ένα τμήμα τη μάχη της ενάντια της κατακτήσης των σημερών ευκαιρίας, τελεία, και να απακολουθήσει το δεύτερο τμήμα που έχει και να αναπτύξει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μητρώου. Η άλλη τροπολογία που θέλουμε ε, και είναι πάλι εδώ να υιοθετηθεί η πρόταση για split vote, είναι η 34. Το πρώτο της ε, τμήμα καλεί τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των διεθνών συνδικών όπως η STCW και η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 να βελτιώσουν και να εξυγχρονίσουν τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης για την περαιτέρω ποιοτική εξέλιξη των ναυτικών σχολών παράλληλα και εκεί να πάει το δεύτερο τμήμα μετά τη συνέχεια που έχει να κάνει με τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων και μπαίνουν ζητήματα ως ελάχιστες οργανικές συνθέσεις που πρέπει να, θεσπιστούν, να θεσπιστούν για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς αλλά πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι μέσα στα πλοία και στους συναφείς κλάδους, ναυπηγεία, λιμάνια, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς παρακολουθούν ε, τη συνεδρίαση και τις αποφάσεις ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να επισημάνω το εξής και να τελειώσω. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στην Ελλάδα πουλήθηκαν την τελευταία 15 ετία τέσσερις φορές. Και ακούστε εδώ το πρωτότυπο. Πού υπάρχει αυτό σε κάποιο κράτος στον κόσμο. Η Group, μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που ελέγχει πάνω από αυτά ναυπηγικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονάδες στο Χάλιμπα, σε μια σειρά κλάδους και τομείς, να έχει έτοιμα τρία υποβρύχια, τρία υποβρύχια, στα, για τα οποία έχει προπληρωθεί ένα μεγάλο ποσό στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, να μην τα δίνει στην ελληνική κυβέρνηση, στην προηγούμενη ή και στην νέα που εκλέχθηκε; γιατί έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα ναυπηγείο ένα στην ε, Γερμανία που κατασκευάζει το υποβρύχιο Πανικολής που έχει σοβαρά προβλήματα. Φτάσαμε δηλαδή εδώ όχι μόνο οικονομικοί όροι να παίρνουν την, ε, το χαρακτήρα του πολέμου, αλλά να μπαίνουμε και σε ουσιαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των κρατών μελών. Νομίζουμε ότι είναι προβλήματα που πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα συνεχίζοντας αυτή την ε, πολιτική θα διωγκωθούν. Πολωνία, Ναυπηγία, Ισπανία, Πορτογαλία, στην ίδια ρότα, στην ίδια κατάσταση. Χρειάζεται πραγματικά ε, να αλλάξει ριζικά αυτή η πολιτική και πιστεύουμε έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Ευχαριστώ ο Αντιπρόεδρος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συντομότατα. Επειδή είναι πολλές οι τροπολογίες που κατέθεσα με τον Βλάστο, θα ήθελα να εξηγήσω. Η έκθεση είναι εξαιρετική. Δεύτερον, ο λόγος ύπαρξης αυτών των τροπολογιών είναι για να μεταφερθεί η προβληματική αυτή των θαλασσίων μεταφορών στη συνολική λογική των μεταφορών. Γιατί υπάρχουν μεν ιδιαιτερότητες στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά πολλές φορές αγνοείται το γενικότερο πλαίσιο. Γι' αυτό ήθελα να ξανασκεφτούμε τις επιπτώσεις του τρόπου αυτού μεταφοράς στο περιβάλλον δεν είναι και τόσο καταστροφικές. Εξάλλου για την έρευνα ανάπτυξη και συμπερίληψη στα δίκτυα γενικότερα οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να θεωρηθούν ως ένας κρίκος της συνολικής αλυσίδας των μεταφορών έτσι ώστε να μπορέσουν να του εφαρμοστούν και τα διάφορα διαρθρωτικά προγράμματα όπως και οι συνδυασμένες μεταφορές. Γι' αυτό οι τροπολογίες αυτές ε, συμπληρώνουν συνήθως την έκθεση αλλά δεν είναι κατά του πνεύματός της. Ευχαριστούμε για την Κομισιόν. Ο κύριος Καραμίτσος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση και την πολύ χρήσιμη συζήτηση που προκάλεσε σήμερα εδώ. Θα επανέλθω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που με ενδιαφέρει και μένα ιδιαίτερα γιατί με εντυπωσίασαν αυτά που είπε ο κύριος Τούσας για την κοινωνική πτυχή του θέματος. Για να αποσαφινιστούν τα πράγματα περαιτέρω, πρέπει να γνωρίζει ο κύριος Τούσας ότι η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής μας δεν αγνοείται, είναι στο πάνω-πάνω των προτεραιοτήτων μας. Είναι κάτι δηλαδή που το θεωρούμε τεράστια σημασίας. Να παραμείνουν γνωστά όλα αυτά και η γνώση να παραμείνει μέσα στην Ευρώπη όχι μόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές, για ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία θέματα που εθίγησαν και από τους ομιλητές. Πρώτον, για το πρόγραμμα συναλλαγών εκπομπών, το λεγόμενο INDS. Πρώτον, πέρυσι, στις 23 Απριλίου μάλιστα, ελήφθη μία απόφαση κοινή από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που καθόριζε ρητά το χρονοδιάγραμμα. Έλεγε πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Θαλασσίων Μεταφορών να καθοριστούν στόχοι. Αυτό εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη και μόνο αν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία μέχρι τις 31 Απριλίου 2011 τότε μόνο η Κομισιόν να κάνει προτάσεις για τις εκπομπές διοξιδίου από τις θαλάσσιες μεταφορές. Άρα αυτό που συμφώνησε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι να προσπαθήσουμε το πρόβλημα να το λύσουμε μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Θαλασσίων Μεταφορών. Και μόνο αν μέχρι το τέλος του 2011 το ξαναλέω δεν υπάρχει συμφωνία τότε μόνο πρέπει η Κομισιόν να προσπαθήσει να το δει περιφερειακά. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πολύ απλός. Πρώτον, εάν δεν καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να μπορεί ο εφοπλιστής να αλλάζει σημαία ή να αλλάζει κατηγορία του πλοίου για να αποφύγει τις ευθύνες του. Και άρα δεν θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός της μείωσης των εκπομπών. Και δεύτερον, σήμερα ήδη ισχύει στην νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια κτλ. Ό,τι ισχύει για αυτά δεν θα μπορεί να ελεγχθεί πια με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό μετά από μεγάλη συζήτηση της μόνιμης αντιπροσωπείας στα τέλη του προηγούμενου χρόνου καταλήξαμε τελικά σε μια δήλωση της Προεδρίας για το πρόγραμμα δράσης μείωση των εκπομπών διοξιδίου από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και η επόμενη τέτοια συζήτηση θα γίνει αυτή την εβδομάδα αν δεν απατώμε. Σας διαβάσω τι λέει το σχετικό κείμενο. Τα ευρωπαϊκά κράτη συμφωνίζουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες να μειώσουν τα κράτη-μέλη τις εκπομπές αερίων με εφέδερμο κρυπίου και έτσι τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν με τη Διεθνή Οργάνωση Θελασσίων Μεταφορών για να μη χωρίς να στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου 2011. Αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Αν δεν προσπαθήσουμε να υπάρξει αυτή η Διεθνή Συμφωνία θα γίνει η στρέβλωση. Έτσι λοιπόν ως Ένωση και ως κάτι μέλη μεμονωμένα πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια στο διεθνές επίπεδο. Τώρα, πέραν από το πρόγραμμα συναλλαγών εκπομπών, υπάρχουν και συζητήσεις για τη δημιουργία ενός, λέει, ταμείου ή διεξέβρεση τεχνικών μέσων για τη μείωση διεθνώς των εκπομπών με εφέδερμο κηπίου. Έπειτα υπάρχει το θέμα των κρατικών επιχορηγήσεων και του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας μάλλον. Είναι σημαντικό μέσα στην τωρινή κρίση να διατηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Μέχρι το 2011 ίσως χρειαστούν ορισμένες αλλαγές, αλλά προς στιγμήν μόνο θετικές επιπτώσεις έχουν υπάρξει. Δεν χάθηκαν πλοία για να που να φύγουν εκτός Ένωσης. Αντίθετα έχουν γίνει αιτήσει για προσθήκη πλοίων από έξω. Αποφύγαμε δηλαδή τουλάχιστον αυτά που έγιναν τη δεκαετία του 80 πολύ outflanking και άρα απώλειες θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Μετά, μετά για τις τροπολογίες. Αν θέλετε μπορώ να τις ξεφυλίσω έτσι στα γρήγορα, στα πεταχτά. Η συμβιβαστική α είναι κάτι που μπορούμε να τη δεχτούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι χρήσιμη. Συμβιβαστική β επίσης νομίζω είναι χρήσιμη. Ίσως θα μπορούσαμε και να την ξεπεράσουμε, αλλά τέλο πάντων είναι αποδεκτή. Μία αποσαφήνιση τώρα. Πρέπει να τονίσουμε στο, για τη συμβιβαστική γάμα ότι πρέπει νομίζουμε να σταματάει μετά από εκεί που λέει το 2011 συμφωνία με τη Διεθνή Οργάνωση Ταλαζίων Μεταφορών. Γιατί υπάρχει ήδη μια οδηγία του 2009 κάθετος 13 που έχει μεταφέρει όλα αυτά σε κοινοτική νομοθεσία. Έχουν συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και εδώ πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τη συμφωνία αυτή γιατί μέχρι τώρα μόνο μία χώρα μέλος την έχει εγκρίνει η χώρα της Προεδρίας και είναι σημαντικό και οι υπόλοιπε να την εγκρίνουν ως το δυνατόν συντομότερο. Μετά για το θέμα του συμβιβασμού Δέλτα και εδώ δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Τη συμβιβαστική ε η πειρατεία είναι κάτι που πολλοί προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Υπάρχει συνεργασία και με μας και με διεθνείς οργανώσεις, με την ε, οργάνωση της Αταλάντας ας πούμε. Εκεί που έχουμε περισσότερες αντιρρήσεις ή μάλλον δεν καταλαβαίνουμε καλά είναι η τροπολογία 28 για τη συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Ναυσιπλοεία στο Ρήνο. Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε μόνο με αυτούς, αλλά και με τις ναϊάδες 2 όπως λέμε, δηλαδή τις νέες προτάσεις συνεργασίας με όλες τις επιτροπές του Δούναβη, του Ρήνου, και οποιασδήποτε άλλες. Uh, είναι σημαντικό νομίζω. Για το Ευρωπαϊκό Μητρό, ναι, αυτό είναι παλιό θέμα και επίπονο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα. Σε αυτό καταλαβαίνουμε τις ιδέες που εκφράζονται. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε στις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχορηγήσεις να υπάρξει τουλάχιστον κάποια εναρμόνιση των εθνικών μητρώων. Τώρα για το Ευρωπαϊκό Μητρό δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Κουμουτσάκο, θέλετε σύντομα να παρέμβετε. Σε συνέχεια του επιχειρήματος που ακούστηκε για την παράγραφο 34 όπου ζητήθηκε split vote ε, προφανώς ο συνάδελφος κύριος Τούσας δεν έχει καταλάβει ότι αυτό το οποίο εισάγεται σε αυτή την παράγραφο ή εμείς δεν το έχουμε εκφράσει καλά είναι ακριβώς για να προστατεύσει κινείται στην δική του λογική και στη δική του κατεύθυνση διότι αν δεν υπήρχε το μίνιμουμ ε, αριθμού πληρώματος μπορεί στα πλαίσια του ανταγωνισμού να μην γινόταν σεβαστό ούτε αυτό το μίνιμουμ επομένως κινούμεθα στη δική του λογική αλλά πέραν αυτού θα ήθελα δύο μικρές επισημάνσεις κύριε Πρόεδρε στην παράγραφο, στη, όσον αφορά την ε, τροπολογία 52 από τους συναδέλφους Βλαστό και Ρικέ, θα ήθελα να πω ότι uh, προτίθεμαι να εισάγω μια ε, προφορική τροπολογία που νομίζω ότι θα έκανε και τον εισηγητή να αντιμετωπίσει θετικά τη συγκεκριμένη τροπολογία. εκεί θα πούμε η, η προφορική τροπολογία θα είναι σαφώς λιγότερο δεσμευτική από την ήδη προταθήσα. Δηλαδή θα κινείται στη λογική του ότι, και το λέω στα αγγλικά, «The sector can contribute to the fight against harmful emissions and climate change» can instead of uh, should or will. Το ΜΕΣ μπορεί να ενεργήσει κατά βλαβερών νεκρών και μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει ιδιαίτερα τις δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις. Σε, σε λιγότερο αυστηρή κατεύθυνση και ελπίζω ότι και ο κύριος Βαντάλεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με αυτή την προφορική τροπολογία. Τέλος, ε, για, την, ε, για την συμβαστική πρόταση D θα ήθελα να πω εκ μέρους του, του EPP ότι θα θέλαμε η η συμβιβαστική αυτή πρόταση να καλύψει και τις τροπολογίες 63 και 64 από τους συναδέλφους του ΙΠΠ Βλαστό και Κούν. Επομένως, η τροπολογία D, στην τροπολογία D να είναι ομπρέλα και για τις ε, τροπολογίες 63 και 64. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουμουτσάκο, δεν ξέρω αν, αν μας είπατε ότι θέλετε να παρουσιάσετε σε, σε αυτά τα σημεία προφορικές τροπολογίες, εάν υπάρχει αντίρρηση μπορούμε να παρουσιάσουμε τις ε, προφορικές τροπολογίες και αν έχουμε το περιεχόμενο των προφορικών τροπολογιών. Τώρα με έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω είναι καινούργιο το αίτημά σας για προφορική, προφορικές τροπολογίες ή παλιό αίτημα για προφορικές τροπολογίες. Να μας φωτίσει ο κύριος Γκρός, ελπίζω. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος παρουσίασε αυτό το οποίο έτσι και αλλιώς θα υποβάλουμε γραπτά στη γραμματεία για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση αύριο στην ψηφοφορία και ότι ο συμβιβασμός καλύπτει και τις δύο τροπολογίες. Διαφορετικά θα είχαμε πρόβλημα στη λίστα, αλλά αύριο το πρωί θα τα εξηγήσουμε. Πολύ ωραία, χαίρομαι λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Βαντάλε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Έχουμε μερικά σημεία που πρέπει να τα εξετάσουμε καλύτερα γιατί άκουσαμε ερωτήσει ε, και σχόλια η 54 δόθηκε από την Επιτροπή μια ιδιαίτερα συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Στην κατάλληλη ψηφοφορία εγώ θα υποδείξω αρνητική ψηφοφορία. Μετά πώς ακούσαμε τον κύριο Καραμίτσο. Μετά το αίτημα Φλακεστάιν που αναφερόταν στην τροπολογία 22 Εκεί γιατί αυτή η συμβαστική τροπολογία υπάρχουν διαφορές πέρα από το σημείο αναφορά στο αν δεν θα πρέπει να υπάρξουν κρατικές επιδοτήσεις εντάξει πάνω σε αυτό αλλά να δούμε τις εξαιρέσεις για να μπορέσει κανείς να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις κρατικές ε, ενισχύσεις. Αλλά στο θέμα αυτό για την αυτιλία δεν θα πρέπει να υπάρχουν, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι σοσιαλιστές. Γι' αυτό ακριβώς η συμβαστική μου η Β είναι καλύτερα, καλύτερη νομίζω από την συμβαστική από την ε, τροπολογία του συναδέλφου. Αυτέ είναι σημαντικέ για μένα τροπολογίε, Πρόεδρο. Και μετά για τον κύριο Φλανκεστάιν, για την τροπολογία 82. Στην τροπολογία 82. Συγγνώμη, 83 διορθώνει ο, ο, ο ζητάει μια προσθήκη του δεύτερου μέρους ή του τρίτου μέρους. Δεν κατάλαβα καλά. Το δεύτερο. Το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος λοιπόν. Αυτό κατάλαβα. Και τα διάφορα αλλιευτικά. Δεν το είχα καταλάβει στην αρχή καλά. Ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν. Φλάκεστάιν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα, πώς θέλετε το θέμα στην 83. Ένα λεπτό στο 83. Στο τέλος προτείνεται, στο, προς το τέλος, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση της πειρατείας. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτά που πολύ σωστά είπαμε προηγουμένως και στις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά εδώ θέλουμε να τονίσουμε ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια αντιμετώπιση, παγκόσμια προσέγγιση. Να μην λείψει αυτό το στοιχείο. Κατά τα άλλα συμφωνούμε με τη συμβαστική τροπολογία. Ωραία. Εντάξει τότε. Στο τρίτο μέρος της τροπολογίας 83 έχω ορισμένε απορίες διότι δεν θα ξέρω, αν, δεν ξέρω αν θα πρέπει σε μια γενική έκθεση να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Δεδομένου το Κοινοβούλιο έχει ιδιοθετήσει μια κοινή θέση επί της πειρατείας, δεν ξέρω αν θα πρέπει να επισέλθουμε σε τόσες λεπτομέρειες. Βεβαίως αν οι ομάδες καταλήξουν σε άλλο συμπέρασμα θα το σεβαστώ, απλώς αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεδομένου ότι μιλάμε για στρατηγικούς στόχους και έτσι γενικά. Και μερικά άλλα σημεία, αλλά πιστεύω ότι πριν ψηφίσουμε αύριο θα έχουμε συγκεράσει τις απόψεις μας. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα είναι η Βαλτική θάλασσα και η στρατηγική της Ένωσης. Κύριο κύριος έχει το λόγο, είναι και εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών πιστεύω ότι θα πρέπει σαφώς να εκφράσουμε την άποψή μας για μια στρατηγική στην περιοχή της Βαλτικής, στην περιφέρεια της Βαλτικής. Είμαι εισηγητής και έχω συγκεντρώσει την προσοχή μου στα θέματα μεταφορών αλλά και στα θέματα τουρισμού, δεδομένου ότι η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη και για την τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν ως και όδης ε, εισηγητές ε, στην ομάδα με πολύ συνεργατικό πνεύμα. Παρουσίασαν λοιπόν τις τροπολογίες τους και ε, είπαν ότι γενικά έχουν μια θετική άποψη. Γι' αυτό ακριβώς και οι τροπολογίες είχαν ένα θετικό πνεύμα και προσπάθησα να τις ενσωματώσω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πέραν της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Αδρυτική και τη Σκανδιναβία και βεβαίως την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Έχουμε υποβάλει δύο συμβιβαστικές τροπολογίες, Γκάνσιαν και Σεμόνοβα, οι οποίες καλύπτουν οι συμβιβαστικές τροπολογίες ακριβώς αυτό το θέμα. Επίσης θέλαμε να τονίσουμε και την σιδηροδρομική διασύνδεση, δηλαδή την διασύνδεση των μεταφορών από τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τρίτων χωρών. Η κυρία Σαβιζάρ και ο κύριος Μαρινέσκου έχουν υποβάλει τροπολογίες για την ενίσχυση προς Ανατολάς μεταφορικής ικανότητος. Εν συνεχεία, επίσης, θέλουμε να διευρυνθούν οι διευρωπαϊκοί άξονες TEN υπαριθμών 1 μέσω Βερολίνου προς τη Δανία και εκεί συμφωνήσαμε σε αυτόν τον άξονα Βέβαια, υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένε πτυχές στις συγκεκριμένες μεταφορές και γι' αυτό ε, παρουσιάστηκαν και οι τροπολογίες του κυρίου Τσίλε στο 2, α, τροπολογία 2 Τσίλε με μια διαφορετική διατύπωση στην ίδια ουσία Ορισμένες ε, τροπολογίες τις οποίες ε, δεν δέχομαι έχουν αρνητικό πρόσημα. Το δικαιολογώ αυτό επειδή έχουν υπερκαλυφθεί ήδη από άλλες τροπολογίες ή καλύπτονται από το κείμενο. Δεν θέλω να επικαλύπτονται οι τομείς των μεταφορών με τον τομέα του τουρισμού. Θέλω να υπάρχει σαφής πολιτική στον κάθε τομέα. Αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι η πλευρά των εκπομπών ε, και των ρήπαντων στις ε, θαλάσσιες μεταφορές, ε, δεδομένου ότι θέλουμε να επεκτείνουμε τους θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους, βεβαίως χρειαζόμαστε έρευνα και ανάπτυξη R&D αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν ταιριάζει ε, στο σημείο που συζητάμε και επίσης η συμπερίληψη τρίτων χωρών. Αυτό έχει παρουσιαστεί ως αίτημα σε αρκετές τροπολογίες. Δεν έχω αντίρρηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η στρατηγική μας στη Βαλτική θάλασσα να τη διατηρήσουμε σε μια συγκεκριμένη γραμμή, δηλαδή να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε επικοδομητικές μεταφορές ε, με σεβασμό προς το περιβάλλον, ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών, συνδυασμό σιδηροδρομικών και θαλασσίων μεταφορών. Μιλήσαμε μόλις για την αυσιπλοεία, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε γενικά τις μεταφορικές ικανότητες προς Ανατολάς ώστε να καλύπτουμε και την περιοχή της Βαλτικής και να μην δεχνάμε και τις οδικές μεταφορές. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες και οι συμβιβασμοί είναι καλοί, είναι θετικοί. Όσον αφορά την πτυχή του τουρισμού, εδώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση της Βαλτικής ε, περιφέρειας ε, με τις ε, γειτονικές χώρες, με την αύξηση του τουρισμού από τις χανζεατικές περιοχές, την ενίσχυση των, του τουρισμού και της ποδηλασίας, της τουριστικής ποδηλασίας 19 τροπολογίες νομίζω δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα και θα υπερψηφιστεί η έκθεση. Ευελπιστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτσάιτης από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για τις εργασίες που έχει κάνει. Συζητήσαμε δελεχώς τη γνωμοδότηση η στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής πρέπει να διαμορφωθεί με μια ευρεία προοπτική Πράγματι, οι ενισχύσεις για τις διάφορες μορφές μεταφορών τονίζονται σε αυτή την έκθεση, συνδρομικές, θαλάσσιες, οδικές και ζητείται η εδραίωση, η ανάπτυξη επαρκών ε, μεταφορών, ε, ασφαλών μεταφορών. Όμως, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία μας ε, που συζητήσαμε και στην ομάδα εργασίας που θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τον τομέα, την περιφέρεια της Βαλτικής. Στόχος μας δεν είναι και η τουριστική και η μεταφορική ανάπτυξη και η ευκολότερη πρόσβαση από τα άλλα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν δεν υποστηρίχθηκε η δική μας πρωτοβουλία. Επίσης θα πρέπει βεβαίως οι καλύτερες προτάσεις των πρασίνων να ληφθούν υπόψη διότι έχουν πολύ καλές ιδέες όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στην, ε, στις υποδομές. Επίσης η χρήση της ηλιακής και ολικής ενέργειας και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να τονιστεί. Πιστεύω ότι εάν εγκρίνουμε 18 από τις 19 τροπολογίες, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης θα αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος, μεγαλύτερο βάρος και έτσι η Επιτροπή Περιφερειών θα, η, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορέσει να παρουσιάσει μια καλύτερη έκθεση. Γι' αυτό πιστεύω, σας παρακαλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και εγώ μιλώ εκ μέρους της κυρίας Σάβησα και πάλι, η οποία ακόμα δεν έχει φτάσει. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Κούν. Βεβαίως ε, είναι μεγάλη απόσταση από την Εσθονία η κυρία Σάβησα είναι παδός τη ποδήλασίας, αλλά δεν νομίζω να έχετε με ποδήλατο και ελπίζω να φτάσει σύντομα. Λοιπόν, η στρατηγική της Βαλτικής Ένωσης είναι η πρώτη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των μακροπεριφερειών και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ε, παραδειγματική και για άλλες μακροπεριφέρειες ώστε να χρησιμοποιηθεί εμπειρία από αυτή την πρώτη στρατηγική. Η Βαλτική θάλασσα είναι σημαντική περιφέρεια, ιδίω στη Βόρεια Ευρώπη και εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερα οι μεταφορές διότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες ελλείψεις. Μόνο με την ανάπτυξη των μεταφορών θα προωθηθεί η εσωτερική αγορά και αυτό αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Βαλτική περιφέρεια χρειάζονται και δημοσιονομικές ενισχύσεις, χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Η Φιλανδία και οι τρεις βαλτικές χώρες δεν είναι σχεδόν καθόλου συνδεδεμένες σιδηροδρομικά και θα πρέπει και τα επιβατικά τρένα αλλά και τα, φορτηγά τρένα να συνδεθούν με άλλες περιοχές, να δημιουργήσουμε μια σιδηροδρομική σύνδεση. Επίσης να ενισχύσουμε την, ε, τις, ναυτιλια, τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως με μορφές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως. Με τον ίδιο, την ίδια κατεύθυνση κινείται και η γνώμη μας για τις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη όπως η Ρωσία η οποία βέβαια συνδέεται με τις βαλτικές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν τις διασυνοριακές σχέσεις ε, να τις λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για το ρόλο των μακροπεριφερειών δεν είναι μόνο η πολιτική συνοχή που μας ενδιαφέρει, αλλά και η διασύνδεση αυτής της περιοχής διεθνώς. Όχι μόνο με γειτονικές χώρες. Ο τουρισμός είναι σημαντικός, βεβαίως θέλουμε να τον ενισχύσουμε, να βελτιωθεί η τουριστική ανάπτυξη μέσα και στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας και γι' αυτό έχουμε τονίσει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού βάσει αυτής της πολιτικής, της μακροπεριφερειακής πολιτικής. Από πλευράς της ομάδας μου πρέπει να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις περισσότερες παρατηρήσεις και με τις τροπολογίες των άλλων ομάδων, με τις περισσότερες. Πιστεύω ότι αύριο θα υπερψηφιστεί, θα υπάρχει και μεγάλη συνένεση απόψεων. Και εγώ εκπροσωπώ την σκιώδη συγγήτριά μας, την κυρία Όρτεν Όκεν, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι σωστή, είναι θετική, προς την σωστή κατεύθυνση. Εδώ και έξι χρόνια που έχουμε τα καινούργια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους ε, έχει αλλάξει η διεθνής ε, ο διεθνής μας προσανατολισμός και έχει ενισχυθεί πολύ περισσότερο η προσανατολάς στρατηγική. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μία μεγάλη γεφύρωση σχέσεων και γι' αυτό ε, πρέπει να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τις μεταφορικές συνδέσεις και μέσω ε, των σκανδιναβικών χωρών παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία στην επανενωμένη Ευρώπη. Η κυρία Μάισεν ήδη ανέφερε τον τουρισμό, σίγουρα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο επειδή είμαστε η αρμόδια επιτροπή, αλλά επειδή η, Λισαβόνα, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ένα άρθρο συγκεκριμένο για τον τουρισμό. Λέει ότι ο τουρισμός θα πρέπει να διαφυλαχθεί και όχι να καταστραφεί όπως έχει γίνει σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτά τα λάθη, τα παθήματα. Μαθήματα, εγώ εάν ζητούσε ένα συγκεκριμένο άρθρο να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη Μεσόγειο, δεν θα το ψήφιζα, ούτε θα πήγαινα για τουρισμό στη Μεσόγειο, όπου έχει επέλθει σχεδόν μια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύξουμε τον καλό και σωστό τουρισμό ε, Πολλές φορές ε, οι χώρες ε, της Βαλτικής αλληλοκατηγορούνται και αλληλοκατηγορούνται και με τις γειτονικές χώρες. Λένε οι Λιθουανοί, οι Πολωνοί δεν μας βοηθάνε γιατί δεν κάνουν και αυτοί κανένα δρόμο, οι Πολωνοί λένε γιατί δεν μας βοηθάνε Είμαι μεν και οι δε. Τέλος πάντων πρέπει εμείς να ενισχύσουμε όλο αυτό το πλαίσιο μεταφορών. Ιδίως ε, Βερολίνο, Ροστόκ, Σκανδιναβία. Αυτό τον άξονα. Όλες οι παράκτιες περιοχές της Μεσογείου θα έχουν καλύτερη προσέγγιση μέσω του άξονα Σκανδιναβία, Ροστόκ, ε, Βερολίνο προς Νότον. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει ε, συνένεση και ευρεία συμφωνία με αυτή την πρόταση και γι' αυτό συμφωνούμε με, με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και ευχαριστώ τον εισηγητή αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές θερμά. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι πάει τα ποδήλατα εγκρίνονται οριστικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κούν που τόσο χρήσιμα μας επέβαλε τις, προτάσεις, τις συμβιβαστικές του προτάσεις. Αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους διότι εγκρίθηκαν οι τροπολογίες μας εδώ. Είμαστε τρεις. Είναι τρεις μάλλον οι τροπολογίες μας και συμφωνώ με όσους είπαν ότι στη Βαλτική πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Σε μεγάλο βαθμό οι ενδιαφερόμενες χώρες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν κανένα τέτοιο σχέδιο ούτε από το Ταμείο Συνοχής ούτε από τους δικούς τους πόρους. Πρέπει λοιπόν η Ένωση να το αναλάβει όταν θα συζητήσουμε τα προγράμματα αυτά γιατί θα μας ε, καταδικάσουν οι λαοί για την καθυστέρηση. Πρέπει να καταλάβετε το πρόβλημά μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούν διότι κατάλαβε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα του του ανταγωνισμού μεταξύ λιμένων της Βαλτικής. Εδώ δεν είναι θέμα που αφορά διαφορές μεταξύ κρατών μελών γιατί καμιά φορά πρόκειται και για λιμάνια στο ίδιο κράτος ή για τις διαφορές που ισχύουν στο Καλίνιγκραντ. Ξέρουμε ότι η Ρωσία δεν σέβεται τα ίδια κριτήρια αποτελεσματικότητας με την Ένωση και το ίδιο ισχύει και για τα περιβαλλοντολογικά. Αν θέλουμε να ληφθούν μέτρα για τη Βαλτική, ενώ τα μέτρα αυτά δεν τα δέχεται η Ρωσία, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί τα μέτρα και τα πρότυπα πρέπει να εγκριθούν διεθνώς ενώ η Ρωσία συνήθως διαφοροποιείται από την πολιτική των χωρών μελών και μεταξύ αυτών των Βαλτικών. Τώρα συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία για μια καλύτερη καλύτερες σχέσεις μεταξύ χωρών και εκτός Ένωσης εξών και η Ρωσία. Η τροπολογία 19 είναι κάτι πολύ σημαντικό διότι προβλέπει 20 εκατομμύρια ευρώ για τη στρατηγική αυτή της Βαλτικής σε διαμεθοριακά προγράμματα, προγράμματα που αφορούν τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και άλλες γειτονικέ χώρες. Και το έγγραφο αυτό νομίζω πρέπει να το εγκρίνουμε διότι πρόκειται όχι μόνο για επενδύσεις αλλά και για κάτι που πρέπει πολιτικά να το στηρίξει η Ένωση. Σας ζητώ λοιπόν να το κατανοήσετε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Κούν. Ο κύριος Κούν ε, συνδύασε πολλές αποκλίνουσες απόψεις πάνω σε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με το έγγραφο αυτό οι μακροπεριφέρειες είναι μια πραγματικότητα καινούρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν κοιτάξουμε αυτές τις ε, περιφέρειες ε, για τις οποίες συζητάμε σήμερα, εκεί θα βρούμε το 1 τρίτο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες επίσης που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 100 εκατομμύρια κάτοικοι που, ε, έχουν, που συνδυάζουν την ευμάρειά τους, την πρόοδό τους με τη θάλασσα. Και δεν καταλαβαίνω και τόσο καλά γιατί αυτός ο διάδρομος μεταφορών να σας πω ότι τώρα τελευταία έχω εκλεγεί και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο διάδρομος μεταφορών, αυτή η διάδρομη μεταφορών είναι τόσο σύντομη. Δεν υπάρχει κανείς διάδρομος που να είναι μακρύς και να μπορεί να συνδέσει το Βερολίνο μέσω της υπόλοιπης Ευρώπης ε, με τη Ρίγα, το Ταλίν, ε, τις πόλεις αυτές, τις πρωτεύουσες αυτές. Δεν υπάρχει ένας άξονας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως ε, συνεργάζεται καλά με την Ρωσία, αλλά για μερικά θέματα τουλάχιστον ε, εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για ορισμένα θέματα οικονομικής φύσεως για μια σωστή ανάπτυξή τους. Εάν ε, δούμε το γιατί εμφανίστηκαν αυτές οι μακροπεριφέρειες, παρατηρούμε σαφώς ότι πρόκειται για λόγους περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και επίσης για οικονομικούς παρόμοιους. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε λοιπόν με αυτά τα σημεία. Αλλά όλα αυτά πώς μπορούν να οργανωθούν πάνω σε ποιους πόρους να βασιστούμε. Δεν διαθέτουμε απάντηση σχετικά. Πρόκειται για κονδύλια του Ταμείου Συνοχής και για ίδιους πόρους των κρατών μελών. Πριν από ένα μήνα στο Ρόστοκ ε, για τη Βαλτική θάλασσα οργανώθηκε μια διάσκεψη και εγώ συμμετείχα εκεί και συζητήσαμε για τα σχετικά θέματα με εκπροσώπους της Επιτροπής, οι οποίοι και εκείνοι συμμετείχαν στο φόρουμ αυτό. Και να σας πω ότι ένας ευρωπαϊκός χάρτης με 5, 6, 10 μακροπεριφέρειες, δεν μπορεί κανένα να τις φανταστεί, χωρίς να, και αν, και αν στη μέση βρίσκεται κάτι που να μην αντιστοιχεί σε μια παρόμοια μακροπεριφέρεια, αν δεν έχουμε φτιάξει κάτι το κατάλληλο, το αντίστοιχο λοιπόν. Κάθε μακροπεριφέρεια χρειάζεται μια σύνδεση οικονομική με τους γύρω και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το εξετάσει λεπτομερέστερα για την πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων. Για την πρόταση στα κείμενα τα οποία εξετάζουμε σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική συνοχής δεν προχωράει ιδιαίτερα, δεν υπάρχει μια κατάλληλη της ε, επεξεργασία. Πάντως ε, κατά γενικό τρόπο το υποστηρίζω αυτό το κείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Κύριε Κίνη, θα θέλατε να απαντήσετε σε ό,τι υπόθηκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που στα βασικά σημεία συμφωνούμε. Πολιτική συνοχής σημαίνει πάντοτε ότι πρέπει να είναι παρούσα η συνοχή των κρατών μελών και η συνεκτική δεσμή. Για να το επιτύχουμε λοιπόν αυτό θα πρέπει οι μεταφορικές οδοί να αναπτυχθούν, να στηριχθούν, διότι είναι αλήθεια όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά πρέπει να μπορούμε να φτάσουν τα προϊόντα και στις χώρες στόχο, στις χώρες όπου θα απολυθούν. Γι' αυτό εμείς ως πολιτικοί επί των μεταφορών πρέπει πάντοτε να έχουμε σαφείς στόχους ενίσχυσης των διευρωπαϊκών δικτύων και δι' για τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να ενισχύσουμε, να διευρύνουμε και να αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και εκεί οι βαλτικές χώρες μπορούν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κ. Μπαλτσούτης το ανέφερε και τον ευχαριστώ. Οι τροπολογίες του 15 και 6 τις έχουμε ήδη ενσωματώσει το, την κοινή μας θέση θα τις, θα τις ε, θα υπάρχουν λοιπόν, θα μετωθούν Όσον αφορά τώρα την ε, ανταγωνιστικότητα των λιμανιών, ο κύριος Τσίλε ήδη μας επέστησε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα το οποίο άπτεται της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε συζητήσει την ανταγωνιστικότητα και στο προηγούμενο θέμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις θαλάσσιες μεταφορές. Βεβαίως, οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας της ναυσιπλοείας και επίσης τους ε, κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Μόνο έτσι μπορούν να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές συνθήκες και θα παρακολουθούμε αυτές τις ε, πολιτικές τους. Ο τουρισμός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη Βαλτική θάλασσα και στις ανατολικές περιφέρειες. Το τονίζουμε ιδιαίτερα. Μεταφορές, ε, ε, επιβατικές μεταφορές, αλλά και τουρισμός. Οδικές, υδροδρομικές, θαλάσσιες. Όταν οι μεταφορές αυτές είναι καλές, τα δίκτυα είναι καλά, αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Η πραγματικότητα των βαλτικών χωρών αναφέρθηκαν από πολλούς, από πολλούς συναδέλφους που προέρχονται από αυτή την περιφέρεια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να συνεννοούνται και οι γειτονικέ χώρες σε διμερή ή τριμερή βάση, ώστε να τα βρούνε. Ένας βασικός στόχος είναι να αναπτύξουμε και λογικά, με συνέπεια, τη χωροταξική πολιτική μας, τη χωροταξία, παραδείγματος χάρη, που θα εγκαταστήσουμε στο μέλλον αιωλικά πάρκα η Βαλτική θάλασσα είναι ε, η ναυσιπλοεία στην Βαλτική θάλασσα είναι πάρα πολύ έντονη, έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές και θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Γι' αυτό σκέφτηκα με πολύ προσοχή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τα με τα σκάφη πιλότους, με τη διευκόλυνση της προσέγγισης και της εξόδου των λιμανιών, ε, με τη βελτίωση της ποιότητας ε, των ε, παραλιών. Πώς θα εξασφαλίσουμε τον τουρισμό αν δεν φτιάξουμε την ποιότητα. Επίσης, η όλη υποδομή των έργων και η συμμετοχή των γειτονικών χωρών σε αυτά τα μεγάλα έργα. Εφόσον εγκρίνουμε ή προωθούμε μεγάλα έργα υποδομής, είτε αφορά ενέργεια, είτε αφορά φυσικό αέριο, ε, από πού θα περάσουν τα δίκτυα, πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων, πώς θα συνεργαστούν οι γειτονικές χώρες και πού θα δώσουμε βάρος στον τουρισμό, ταυτόχρονα επισημένοντας τις περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και φυσικού ενδιαφέροντος. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε ανάπτυξη δικτύων, ενίσχυση επενδύσεων και μεγάλων έργων και προστασία του τουρισμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για την περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας ε, είναι πολύ σημαντική, πρέπει να προωθήσουμε την άποψή μας και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και πολλές άλλες περιφέρειες της Ευρώπης να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο όπως είπαμε μαζί με τις υπόλοιπες εκθέσεις. Επόμενο σημείο η δική μου έκθεση εξέταση τροπολογιών μεταφερόμενος εξοπλισμός υποπίεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα αρχίσουν, πρόκειται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το θέμα και εγώ έχω υποβάλει μόνο μία τροπολογιούλα, κανείς άλλος δεν υπέβαλε άλλη. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Η πρόσθετη λοιπόν τροπολογία που προϋποβάλλω λαμβάνει υπόψη της τη θέση του Συμβουλίου και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας που λέει ότι πρέπει να γίνει σε σενή συνεργασία με εθνικά σώματα Τώρα με βάση τη συμφωνία αυτή με το Συμβούλιο για τη διατύπωση για αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα να πω ότι θα υποβάλω προφορικές τροπολογίες που θα συμπεριλαμβάνουν τη συμβιβαστική διατύπωση για τις λεγόμενες delegated acts. Οι προφορικές αυτές τροπολογίες που θα υποβάλω αναφέρουν την συμπεφωνημένη ορολογία και τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί. Θα αναφέρουν δε ρητά ότι η συμπεφωνημένη ορολογία δεν αποτελεί προηγούμενο και για το μέλλον. Είναι απλώς κάτι το προσωρινό ώσπου να καταλήξει το Κοινοβούλιο τελικά στη θέση του στη Θεσμική Επιτροπή. Σας είχα ξαναπεί ότι η οδηγία αυτή, η προτινόμενη οδηγία, είναι μια αναθεώρηση για να απλοποιήσει την ισχύουσα και να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τη μεταφορά αντικειμένων υποπίεση. Πιστεύω ότι όταν εγκριθεί θα αυξηθεί όντως, το, θα διατηρηθεί τουλάχιστον το επίπεδο ασφαλείας που υπάρχει για τη μεταφορά αντικειμένων υποποίηση. Η αναθεώρηση αυτή κατέστη απαραίτητη λόγω διαφορών που σημειώθηκαν στη νομοθεσία για άλλα θέματα και λόγω διεθνών συμφωνιών που είχαν συναυθεί εντωμεταξύ. Και έτσι καταλήξαμε σε αντιφάσεις. Οι τροπολογίες που συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου ζητούν μια αποσαφήνιση των διαδικασιών, ζητούν από την Κομισιόν να μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές προς την πρακτική εφαρμογή των ε, προτάσεων και μια επιβεβαίωση ότι δεν χρειάζεται νέα πιστοποίηση συμβατότητας εάν έχει αυτή δοθεί από τον αρχικό παρασκευαστή το Συμβούλιο δέχτηκε τις αλλαγές αυτές και πράγμα για το οποίο χαίρομαι ιδιαίτερος. Ελπίζω αύριο να εγκρίνουμε τις προφορικές τροπολογίες που έχω υποβάλει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και έτσι το θέμα να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για πρώτη ανάγνωση. Όπως είπε το Συμβούλιο, θα μπορούσε να δεχτεί τις τροπολογίες αυτές. Τώρα το ιστορικό είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κοντέινερ για υποπίεση αέρια και ο στόχος είναι η ασφαλέστερη δυνατή μεταφορά τους μεταξύ των χωρών μελών χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη άδεια και επιστοποίηση και κάθε περίπτωση από κάθε κράτος εφόσον βέβαια υπάρχει σωστή πιστοποίηση από τον παρασκευαστή. Ξέρουμε ότι το θέμα είναι τεχνικό, δεν είναι πρόθεση κανενός να αλλάξει για όντας το περιεχόμενο άρδιν της οδηγίας, αλλά απλώς να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Και όπως σας είπα πριν, αυτό έγινε, κατέστη απαραίτητο γιατί είχαν αλλάξει άλλα νομοθετήματα και γιατί συνάφη, υπήρχαν διεθνεί συμφωνίες που άλλαξαν τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν οι τροπολογίες που έβαλα να αποσαφηνίσουν τους ορισμούς και επειδή ζητώ κατευθυντήριο γραμμές από την Κομισιόν για την πρακτική εφαρμογή των προτάσεων αυτών και αποσαφήνιση ότι δεν θα είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση και από κάθε κράτος η νέα πιστοποίηση, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση του κατασκευαστή, ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε όλα αυτά, τις τροπολογίες που υπέβαλα, τις προφορικές και τις γραπτές, πράγμα το οποίο θα μας δώσει καλύτερη ευκαιρία να κάνουμε γρηγορότερα μια πρώτη ανάγνωση, που, γιατί όπως είπα και το Συμβούλιο δέχεται τις προτάσεις μου αυτές. Και τώρα ο κύριος Ρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξ του ΕΛΚ θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε την τροπολογία σας. Πιστεύω ότι η τεχνική προσαρμογή είχε οριμάσει και ήρθε η κατάλληλη στιγμή να το ψηφίσουμε διότι έχει και προστιθέμενη αξία στο, διασυνοριακές μεταφορές όπου θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και όχι να μειώσουμε τα πρότυπα, τα standards. Για μένα, για την περιοχή από όπου κατάγομαι, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Ειδικά αυτά που είπατε για, την το νομοθετικό πλαίσιο και σε αυτό σας υποστηρίζουμε και γενικά πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε εξαιρετικά σύντομα. Ε, το ΕΛΤ σας υποστηρίζει σε όλες σας τις τροπολογίες που είναι και πάρα πολύ λίγες <laughs> βεβαίως σε σχέση με τα άλλα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Εδώ έχουμε, πιστεύω, πολύ συντριπτική συνένεση. Δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε τίποτα, απλώς να εξαλείψουμε παρανοήσεις και κακές ερμηνείες. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια μεταφορών επικίνδυνων ε, προϊόντων και εξοπλισμού υποποίηση. Είπατε ότι υπάρχει συνένεση απόψεων για το τι πρέπει να πράξουμε και έτσι θα ακολουθήσουμε τη δική σας τη γραμμή αυτή τη και αυτή τη φορά. Επίσης να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω κύριε Σίμψον ε, για την εργασία σας ως εισηγητού είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο αυτή η σαμφίνια την οποία προσφέρεται διότι δεν υπάρχει αυτή η σαφήνεια από απόψεως ε, συνθήκης της Λισαβόνας και γι' αυτό πιστεύω ότι το σχέδιό σας αποσαφηνίζει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία πρέπει να περιληφθούν ε, και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται. Γι' αυτό γενικά συμφωνούμε με όλο το περιεχόμενο της ε, γνωμοδότησής, της ε, γνωμοδότησής σας και θα το δείτε αυτό αύριο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κράμερ, εάν, εφόσον έχεις την υποστήριξη και του ΕΛ και των φιλελευθέρων και τη δική μας, θα πρέπει να σκεφτείς μήπως έχεις κάνει κάτι λάθος. Λοιπόν, χαιρόμαστε για την ψηφοφορία αύριο και υποστηρίζουμε. Ο πρόεδρος προσπάθησα να βάλω κάπου τα ποδήλατα μέσα στο, στο θέμα του εξοπλισμού υποπίεση. Αλλά δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα. Ε, μπορώ να οδηγήσω το ποδήλατό μου, λέει ο κύριος Κούνες, στις συνδρομικές γραμμές, άμα χρειαστεί. Λοιπόν, το δύναμό μου σημείο είναι αυτό, λέει ο πρόεδρος. Ακούστε, εμείς εμείς ε, δεν θέλαμε να πούμε ότι δεν θέλαμε να σας υποστηρίξουμε. Όχι, το αντίθετο. 100% σας υποστηρίζουμε και σας ευχόμαστε το καλύτερο. Εμείς θα σας υποστηρίξουμε, λέει ο κύριος Ζήλε, γιατί η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και επειδή ο τρόπος που χειριστήκατε το όλο θέμα είναι εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κ. Πασκουάλε από την Κομισιόν. Εάν και εσείς με υποστηρίζετε, η θέση μου είναι δυσχερής. Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ σας υποστηρίζω και σας ευχαριστώ για την πολύ επικοδοματική σας θέση, έτσι ώστε μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε επί του κειμένου σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την ε, ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για τον οικονομικό τομέα. Αύριο θα ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος, αύριο το πρωί σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, σοβαρά τώρα, ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας, ευχαριστώ. Ωραία, πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την, τις εργασίες της Επιτροπής μας για το απόγευμα σήμερα και έχουμε τους συντονιστές στις 5.30. Αν είναι όλοι οι συντονιστές εδώ, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και να αρχίσουμε μετά το συντομότερο. Ευχαριστώ.